Η, πρόεδρο πρόεδρος Γκρέσλε. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Κυρίσω την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού για θέμα αρμοδιοτήτων ε, ελέγχου. Έχουμε αφιερώσει το σημερινό απόγευμα στις χώρες του Δυτικού, των Δυτικών Βαλκανίων και γι' αυτό καλωσορίζω τους συναδέλφους από Βοσνία Ζεγοβίνη, Αλβανία, από την Φύρομ, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και την Σερβία. Καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε για την παρουσία σας εδώ. Θα περάσουμε μαζί το σημερινό απόγευμα, ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες, αν μου επιτρέπετε. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο, σας παρακαλώ, χρησιμοποιήστε το έντυπο που σας δείχνω. για να μην υπάρξει καμία δυσκολία ε, λόγω των ε, διαφορετικών προελεύσεων κλπ. Ε, σας παρακαλώ να τηρήσετε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 29 τακτικά και 21 αναπληρωματικά μέλη. Συνεδριάσαμε ήδη σήμερα το πρωί και θα ήθελα να αρχίσουμε την απογευματινή συνεδρίαση με παρουσίαση των δικών μας καθηκόντων και του δικού μας τρόπου εργασίας. Στην συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα, δηλαδή η χορήγηση απαλλαγής για τον προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμούς και δαπάνες στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό που είναι της τάξης των 160 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καθήκον της δικής μας Επιτροπής είναι η σύνταξη της σχετικής έκθεσης για την απαλλαγή. Έχουμε δηλαδή τον τρέχοντα προπολογισμό και τον προπολογισμό του επομένου έτου, τον οποίο συντάσσουμε, καθώ και την εκτέλεση του προπολογισμού στο τρέχον έτο και στο προηγούμενο, τα οποία όμω έχουμε χωρίσει σε δύο διαφορετικέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Αυτό ίσω φανεί στι χώρε μέλη κάπω ε, ασυνήθιστο, ο χωρισμό αυτό. Αλλά κάθε χρόνο εκτελούμε τα καθήκοντα αυτά. Είμαι μέλο τη παρούση επιτροπή εδώ και 15 χρόνια. Και όσο περισσότερο εξετάζω την κατάσταση αυτή, τόσο καλύτερο μου φαίνεται το σύστημα αυτό του χωρισμού των αρμοδιοτήτων, διότι θεωρώ ότι όλοι ως βουλευτές οφείλουμε να φροντίζουμε, να διερωτώμεθα και να ερωτούμε ε, πού δαπανώνται τα χρήματα ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. ενώ τα μέλη ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμών κάνουν αγώνα για να επιτύχουν ας πούμε ένα έξτρα κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ, εμείς μετά καλούμεθα δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού να δούμε πού πήγαν τα χρήματα αυτά, πώς εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός. Και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στου ευρωβουλευτές σε αυτή την δραστηριότητα. Εν προκειμένου ασχοληθήκαμε και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, επισκεφτήκαμε πρόσφατα την Αλβανία, έχουμε προγραμματίσει και άλλες επισκέψεις στις ε, χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνεργασία μαζί σας. Η Επιτροπή μας ολόκληρο τον χρόνο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ασχολείται με τον προϋπολογισμό και την εκτέλεσή του. Προχωρούμε τώρα στις εργασίες της απαλλαγής του 2016 και ε, έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια αυτή και προχωρούμε τώρα στο 2017. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 10 θεσμικά όργανα, το μεγαλύτερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή Περιφερειών, εντεταλμένο ε, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Αυτά είναι τα 10 βασικά, βασικά θεσμικά όργανα, τα οποία όλα έχουν δικό του διαχειριστικό προπολογισμό. Και έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειριστικό προϋπολογισμό με προγράμματα, στον οποίο αφιερώνουμε μέγα μέρος των εργασιών μας. Αλλά ασχολούμαστε και με όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, τα οποία όπως εξής είναι 10 στον αριθμό. Έχουμε και 36 αποκεντρωμένους οργανισμούς, 7 joint undertakings, δηλαδή προγράμματα ε, ΣΔΙΤ, των οποίων τους προϋπολογισμούς επίσης ελέγχομαι και τι γίνεται δηλαδή με τα ε, σχετικά κονδύλια, πού πηγαίνουν τα σχετικά κονδύλια. Αυτά αποτελούν το κύριο μέρος των εργασιών μας. Για, μέσα στα πλαίσια των εργασιών αυτών διεξάγουμε ακροάσεις, συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο στέκεται στο πλευρό μας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγει τις εργασίες αυτές επίσης με εντολή από την συνθήκη και για κάθε χρόνο θεσπίζει ποσοστά σφάλματος για όλους τους προϋπολογισμούς. Δηλαδή ασχολούνται να δουν ποιο μέρος έχει δαπανηθεί παρατύπως. Αυτά είναι σφάλματα. Τα ποσοστά αυτά σφαλμάτων θα πρέπει δυνατόν να, να κρατιούνται στο κάτω του 2%. Συνήθως είναι 2 με 5%. Όταν άρχισα εγώ εδώ στα διορθωτικά ταμεία διαπιστώνονταν σφάλματα τη τάξη του 12%. Τώρα έχουμε κατέβει κάτω από τα 5%. Δηλαδή με την μακρά ε, και μακρόχρονη παρατήρηση, με υποβολή συστάσεων και ούτω καθεξή και με άλλα μέτρα έχουμε επιτύχει σημαντική βελτίωση. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή που συνεδριάζουμε συχνότερα, μέχρι τώρα 102 φορέ στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και έχουμε ψηφίσει πάνω από 250 εκθέσει στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και 35 γνωμοδοτήσεις για διάφορα επιμέρους θέματα κάθε χρόνο. Διεξάγουμε τέσσερις αποστολές, τρει σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία εκτός, διότι βέβαια ενδιαφερόμαστε και για τις δαπάνε της Ευρωπαϊκής επιτροπή σε τρίτες χώρε, καθώ και για τι δράσει τη Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνουμε άποψη και έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να οργανώσουμε και ακροάσεις ή εργαστήρια, να αναθέσουμε μελέτες, έρευνες, πράγμα το οποίο κάνουμε, 19 μελέτες για διάφορες, έως τώρα για διάφορους ε, τομείς των ευρωπαϊκών δαπανών. Η βάση των εργασιών μας είναι ο δημοσιονομικός κανονισμός που διέπει τον τρόπο διαμόρφωσης των δαπανών και αυτό είναι σημαντικό για όλους όσοι παίρνουν στα χέρια τους δημόσια ευρωπαϊκά χρήματα. Και αυτό σημαίνει ότι τα όσα κάνουμε εμείς εδώ σήμερα είναι βασισμένα στο νόμο, αλλά γίνεται και μετά από την αντίληψη που έχουμε εμείς για προβλήματα και αυτά που μας τίθεται υπόψη από το ελεγκτικό συνέδριο. Εκτός αυτού είμαστε αρμόδιοι και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου εναλλακτικά με την Επιτροπή Οικονομικών διεξάγουμε ελέγχους για τις δαπάνες της τράπεζας αυτής και για τα αποτελέσματα που υποβάλλει. Ελέγχουμε την τράπεζα στην βάση εκθέσεων και ετησίων εκθέσεων. Είμαστε επίσης αρμόδιοι για την καταπολέμηση απατών συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Απατών Όλαφ και εκτός αυτού είμαστε αρμόδιοι και για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, για τον διορισμό των μελών του, που προτείνονται από τις χώρες μέλη και αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί θα αντιληφθείτε για ποιο λόγο θεωρούμε ότι το έργο μα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε εδώ στο πραγματικό μηχανοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμαστε επί προβλημάτων και ε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε το τι δεν λειτουργεί. Θεωρώ ω καθήκον μας να κάνουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όλα αυτά τα περιλαμβάνουμε σε μια έκθεση, ετήσια έκθεση απαλλαγής. Ο κύριος Τσέλερ, που είναι εισηγητής για την απαλλαγή του 2016, θα λάβει αργότερα το λόγο για να εξηγήσει περισσότερο τις εργασίες μας. Κάθε ένα από τους 36 αποκεντρωμένους οργανισμούς λαμβάνει έκθεση για τα πεπραγμένα του προπολογισμού. ώστε κάθε χρόνο έχουμε συνολικά 52 εκθέσεις. Έχουμε και τις 57 ε, ΣΔΙΤ, δηλαδή συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που ελέγχουμε. Επίσης, αυτά αποτελούν το βασικό μέρος των εργασιών μας. Οι εκθέσεις συντάσσονται πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτικά από έναν εισηγητή. Πρόκειται για αρχή η οποία έχει υιοθετηθεί από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, γιατί έτσι την γνωρίζω και από εκεί, και οι εκθέσει αυτέ κατανέμονται στου εισηγητέ σύμφωνα με την αριθμητική δύναμη των πολιτικών ομάδων. Ο εισηγητή είναι κατά βάση ο υπεύθυνο για να συνοδεύσει μέσα από όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία την έκθεση. Θα κληθούν και οι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ να συντάξουν γνωμοδοτήσει, οι οποίε λαμβάνονται εν τέλει υπόψη στην σύνταξη τελική εκθέσεω. Γι' αυτό άλλωστε και οι εκθέσει φέρουν πάντοτε το όνομα του αρμόδιου εισηγητού. Τώρα ε, σας κοιτάζω για να μου πείτε αν έχω λησμονήσει κάτι, να εξηγήσω. Ε, στην Επιτροπή μας συμμετέχουν μέλη από 7 πολιτικές ομάδες. Κάθε πολιτική ομάδα διορίζει έναν εκπρόσωπο και εγώ σε συνεργασία με τους εκπροσώπους συντάσσουμε το θεματολόγιο, ποιες μελέτες θα ανατεθούν, πού θα γίνουν διάφορες αποστολές, σε ποιες χώρες, ποιος θα συμμετάσχει στις αποστολές, όλα αυτά είναι οργανωτικά θέματα. Εκ δεξιών μου είναι τα πρόσωπα της γραμματείας, που είναι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποστηρίζουν την εργασία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και αριστερά μου οι αντιπρόεδροι, εν προκειμένου η κυρία Ντλαβάζοβα από ε, αντιπρόεδρος, ο κύριο Τάραντ από άλλη πολιτική ομάδα, υπάρχουν ε, αντιπρόεδροι από όλες τις πολιτικές ομάδες, εγώ προσωπικά είμαι από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Το σύστημα του διορισμού του Προέδρου της κοινοβουλευτική Επιτροπής εξαρτάται πάλι από την αριθμητική δύναμη των πολιτικών ομάδων. Ο Πρόεδρος διορίζεται για δυόμιση χρόνια, δηλαδή το μισό της κοινοβουλευτικής θητείας αυτά σε, στην βάση ενός υποδείγματος που όπως λέω έχει πάλι να κάνει με την αριθμητική δύναμη των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Υπάρχουν 23 συνολικά κοινοβουλευτικές επιτροπές και 751 ευρωβουλευτές. Στις 29 Μαρτίου, ως γνωρίζετε, του 2019 θα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τότε θα μείνουμε μόνο 705 προβλεφτές. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην δύναμη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν είναι πάντοτε τόσο δημοφιλής, διότι πρώτον έχει πάρα πολλή δουλειά, λαμβάνουμε πλήθος εγγράφων, χρειάζεται να δουλεύουμε και να διαβάζουμε πολύ και βέβαια χρειάζεται τα θέματα διαρκή παρακολούθηση. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε εδώ την Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση Ανατολική Ευρώπη από το Λονδίνο και ασχοληθήκαμε με τις χρηματοδοτήσει της Ευρωπαϊκή Ένωσης για θέματα αντιμετώπισης της πυρηνικής ασφάλειας, των προβλημάτων πυρηνικής ασφάλειας. Όπως για παράδειγμα μετά από την καταστροφή στο Τσερνομπίλ. Το ίδιο το Τσερνομπίλ Επίση, βοήθειε που χορηγούμε σε χώρε για, την, ε, για την απομάκρυνση ας πούμε αναλωμένων καυσίμων από παροπλισμένα ε, ρωσικά υποβρύχια. Αυτά κρατάνε χρόνια πολλά οι δραστηριότητες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει επίσης την πάυση λειτουργίας πυρηνικών σταθμών σε Σλοβακία και σε άλλες χώρες, τρεις συνολικά, που είναι παλιού σοβιετικού τύπου και χορηγούμε επιχορηγήσεις για να πάυσει η λειτουργία τους. Έχουμε μεταβεί επιτόπου, έχουμε δει τι γίνεται, έχουμε εξετάσει πώς γίνονται οι ε, προκηρύξεις των έργων, ποια προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν, ποιες καθυστερήσεις, ώστε να έχουμε απόλυτα ξεκάθαρη εικόνα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα πράγματα αυτά και δεν ικανοποιούμεθα βέβαια από τις πρώτες δηλώσεις που λαμβάνουμε σχετικά, αλλά διερευνούμε το θέμα σε βάθος. Μαρτίνα, στρέφομαι στην Αντιπρόεδρο κυρία Τζαβάλοβα. Έχετε άλλε παρατηρήσεις εσείς? Καλησπέρα, καλό σας απόγευμα. Η επιτυχία κάθε επιτροπής εξαρτάται από την ε, πρόεδρο ή τον πρόεδρο. Και μπορώ να σας πω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή ε, πρόεδρο και είπε ότι δεν ε, είναι η αγαπημένη επιτροπή αυτή των βουλευτών γιατί χρειάζεται πολύ μελέτη και πολύ διάβασμα και όταν θα μπούμε σε διάφορες διαδικασίες περί απαλλαγής θα το καταλάβετε αλλά ε, εμείς παίζουμε τη δυνατά μας για να τα καταφέρουμε στο κοινοβούλιο. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχω πληρώσει την αντιπρόεδρό μου για να πει τα καλά λόγια. Λέει η κυρία Γκρέσλε Υπάρχουν δύο σχέδια της αρχής του προπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάσσει τον προπολογισμό και βεβαίως και το Συμβούλιο ε, των Υπουργών. Για την απαλλαγή είμαστε εμείς αρμόδιοι ως δεύτερο όργανο. Οι χώρες μέλη υποβάλλουν πρόταση, εάν θα πρέπει δηλαδή να χορηγήσουμε την απαλλαγή όχι. Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο των Υπουργών των Χώρων Μελών, δυστυχώς ξαναλέω, δεν ενδιαφέρεται, δεν εγκύπτει ας πούμε τόσο εντατικά στην διερεύνηση του τι έχουν επιτύχει τα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί, αυτά τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς, ωστόσο που ασχολούμεθα περισσότερο, καμιά φορά ασκούμε και κριτική για τα επιτεύγματα. Και έχουμε αρχίσει τώρα και τη συγκριτική μελέτη μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών. Θεωρώ ότι είναι σημαντική η μέθοδος αυτή, να έχουμε δηλαδή κάποια benchmark, κάποια ορόσημα, κάποιου δείκτες επίδοση που να τους ανακοινώνουμε μετά και στι χώρες μέλη για να γνωρίζουν που βρίσκονται. Οι δείκτες αυτοί είναι για παράδειγμα το ΑΕΠ, είναι οι δείκτες τη ανεργία Για το ζήτημα τι επιτυγχάνουμε, με τα 40 δισεκατομμύρια των δαπανών τη κοινή αγροτική πολιτική. Τι επιτυχάνουμε. Με τα δισεκατομμύρια που δαπανώνται για τα διαρθωτικά ταμεία κάθε χρόνο. Πού καταλήγουν, τι επιτυχάνουμε. Χρειαζόμαστε, όπω είπα, δείκτε, benchmark για να γνωρίζουμε και να γνωρίζουν και οι χώρε μέλη πού βρισκόμαστε και πού βρίσκονται και οι ίδιε στη σειρά. Αυτό σίγουρα θα ενδιαφέρει και τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Η Επιτροπή μας αρνήθηκε την χορήγηση απαλλαγή στο προϋπολογισμό της Κομισιόν το 1999 και τελικώς αυτό απέληξε σε παρέτηση ολόκληρη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι σημαντικό ιστορικό ορόσημο, διότι έκτοτε έχουν καταβάλει όλες οι προσπάθειες να αποφύγουν την επανάληψη τέτοιου επεισοδίου. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι λοιπόν πολύ καλύτερα συντεταγμένο έκτοτε. Θεωρούμε ότι ο ρόλο μα είναι επικοδομητικός οφείλει ε, να υποδεικνύει τα σφάλματα έγκαιρα ώστε να μπορούν να διορθωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχουμε κανένα σκοπό να επικρίνουμε κανέναν ως αυτό σκοπό. Διαπιστώνουμε σφάλματα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα σφάλματα να διορθώνονται. Και αυτό για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για την ώρα ε, δεν θα ήθελα να σας διηγηθώ τίποτε περισσότερο για τις δικές μας αρμοδιότητες και εργασίες. Μπορεί να προκύψουν άλλα τέτοια θέματα στη διάρκεια της συζητήσεως. Αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως. Αν δεν έχετε, να δώσω το λόγο στον κύριο Τσέλερ για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Αν έχετε ερωτήσεις, ξαναλέω, αλλά δεν βλέπω κανέναν να επιθυμεί να ε, θέσει ερώτηση. Ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τσέλερ. Είναι μεγάλη η χαρά μου που βλέπω τόσες και τόσους πολλούς συναδέλφους από τα ε, φύλλα κοινοβούλια, τους οποίους υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, για τα βασικά τώρα, για ποιο, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί ο έλεγχος του προϋπολογισμού και τι οφείλει να κάνει. Τα εξήγησε αυτά λίγο πολύ η Πρόεδρός μας. Είχα την τιμή τα τελευταία τρία χρόνια να ασχοληθώ εντατικά με την χορήγηση απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2014 ως εισηγητής της πολιτικής μου ομάδας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δηλαδή, για τα έτη 2015-2016, ως κοινοβουλευτικός εισηγητής από κοινού με τους εισηγητές των επιμέρους πολιτικών ομάδων που συνεργάστηκαν μαζί μου. Το δίκαιο του προϋπολογισμού είναι το κυρίαρχο δικαίωμα του κάθε κοινοβουλίου. Την απόφαση σχετικά με το κοινοβούλιο λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό, αυτή η απόφαση αποτελεί την βάση για οποιασδήποτε παραπέρα δραστηριότητες του δημοκρατικού μας οργάνου. Είναι σημαντικό βεβαίως να δει κανείς οι στόχοι τους οποίους έχουμε διατυπώσει και τους οποίους επιθυμούμε να επιτύχουμε μέσω του προϋπολογισμού, εάν όντως επιτυγχάνονται και εάν στην προσπάθεια αυτή οι κανόνες εκτέλεσης του προϋπολογισμού έχουν πράγματι τηρηθεί. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το καθήκον πρώτα-πρώτα του, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Στην προσπάθεια αυτή μας βοηθούν οι αιτήσεις εκθέσεις των διαφόρων γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, που λογοδοτούν για τις δραστηριότητές τους, μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού έτους, αλλά μια σημαντική βάση για μας αποτελούν βέβαια οι αιτήσει εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που με τη βοήθεια των συνεργατών του έχει τη δυνατότητα να ελέγχει επιτόπου και σε εντατικό βαθμό την εκτέλεση της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Ο σημαντικότερος εταίρος λοιπόν για μας είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο και πέρα από αυτά, εκτός δηλαδή από την ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εγκύπτει και σε θέματα ειδικά ανατομέα και μας υποβάλλει ειδικά ανατομέα ειδικέ εκθέσεις για επιμέρους έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν σχέση και ενδιαφέρον για τον προϋπολογισμό και αυτό αποτελεί επίσης πηγή για τις δικές μας δραστηριότητες. Γιατί χρειαζόμαστε τις επαφές ιδίως τώρα με τα εθνικά κοινοβούλια ή ακόμα περισσότερο μέχρι και τις περιφέρειες των χωρών μελών. Σε πολλούς τομείς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε στην διαδικασία επιμερισμένης διαχείρισης. Δηλαδή οι στόχοι τίθενται ή μάλλον προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνονται από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο που είναι οι δύο, τα δύο θεσμικά όργανα τα οποία συναποφασίζουν. Εγκρίνονται λοιπόν εφόσον επιτύχουν την συμφωνία και των Ευρωβουλευτών και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων στο Συμβούλιο Υπουργών και μετά περνά το όλον στην εφαρμογή, στην εκτέλεση, την οποία αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. που είναι πλέον άμεση αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περισσότερα, όπω η διαφορετικά ταμεία πολιτική της συνοχής, εξακολουθούν να βρίσκονται στην επιμερισμένη διαχείριση. Δηλαδή, άμεσα για την εκτέλεση του προπολογισμού για την εφαρμογή, αν θέλετε, την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από χρήματα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, άμεσα υπεύθυνε είναι οι χώρες μέλη. Ή εκεί όπου ε, ισχύει η αρχή της περιφερειακής διαχείρισης, όπως σε μεγάλο μέρος των διαρθρωτικών ταμείων, είναι υπεύθυνοι οι περιφερειακοί άρχοντες. Συχνά, συχνά επίσης, όταν υπάρχει κοινή χρηματοδότηση, δηλαδή συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών χρημάτων με εθνικούς πόρους, από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ή όπου συμπληρώνονται, όπου αυτή η δυνατότητα υπάρχει, και από περιφέρειες, οι οποίες φέρουν δικό τους βαθμό ευθύνης και μπορούν να συμβάλλουν με δικά τους χρήματα, έχουμε ειδικού κανόνες ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, που ελέγχουν τους δικαιούχους των τελικών πληρωμών. Για τους επιτόπου ελέγχους λοιπόν, αυτοί γίνονται από τις χώρες μέλη και από τα θεσμικά τους όργανα που έχουν για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εκτέλεση των προβλεπόμενων προγραμμάτων και έργων. Από το ελεγκτικό συνέδριο γίνονται βέβαια δειγματοληπτικοί έλεγχοι, διότι είναι μεγάλος ο αριθμός άνω των 10.000 έργων και δεν μπορεί το ελεγκτικό συνέδριο να τα ερευνήσει όλα. Υπάρχουν μέθοδοι όμως για δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι επιτρέπουν να διαπιστώνεται κατά πόσον τα έργα και προγράμματα έχουν εκτελεστεί με τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό ή αν έχουν σημειωθεί σφάλματα, παρατυπίες είτε των δικαιούχων είτε των διοικήσεων. Εκεί υπολογίζεται το ποσοστό σφάλματος. Ως στόχος εδώ από την πλευρά των θεσμικών οργάνων έχει μπει το ποσοστό σφάλματος κατά των όριων να μην υπερβαίνει το 2%. να μην υπερβαίνει λοιπόν το σφάλμα, το ποσοστό αυτό. Κάτω από το 2% θεωρούμε ότι η δουλειά έχει γίνει σχεδόν άψογα. Για το άνω του 2% θεωρούμε ότι απαιτείται διόρθωση, η οποία θα πρέπει να απολύξει σε εντατικότερο έλεγχο της εκτέλεσης των προγραμμάτων ή και έργων και αν διαπιστωθεί ότι κονδύλια έχουν γίνει ίσως και αντικείμενο κατάχρησης. Και δηλαδή όχι απλώς πρόκειται για σφάλμα, αλλά ενδεχομένως και παρατυπίες. Ή και απάθες. Τότε βέβαια αυτά διώκονται και επομένως πρέπει να εμπλακούν πλέον αρχές όπως η, ο φορεύς, ο οργανισμός καταπολέμησης των απατών. Όλαφ ή εάν δεν έχουν δαπανηθεί σωστά τα κονδύλια θα πρέπει εν τέλει οι χώρες μέλη να αποδώσουν τα εισπραχθέντα. Αυτά όλα είναι μέσα στα πλαίσια της εκτέλεσης του ελέγχου του προϋπολισμού και οι ελεγκτές του προϋπολισμού έχουν τη δυνατότητα στην βάση των γραπτών ετήσιων εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θέσουν γραπτός ερωτήσεις προς τους επιτρόπους, ερωτήσεις οι οποίες θα απαντηθούν και να οργανωθούν και ακροματικές διαδικασίες στα πλαίσια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, όπου προσέρχονται γενικοί διευθυντέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ενδεχομένω και ο ίδιο ο αρμόδιο επίτροπο κάθε φορά προσωπικά για να δώσουν απαντήσει προφορικά. Για μας σημαντικό είναι να προσέρχεται ο αρμόδιος για τον προπολογισμό επίτροπος, εκπροσωπώντας και το συλλογικό όργανο των επιτρόπων. Για το ζήτημα τώρα της επιμερισμένης διαχείρισης, είναι ένα θέμα όπου διαπιστώνουμε πάντα το μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων. Όπου δηλαδή υπάρχουν, υπάρχει συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρήματα και από εθνικά. Όπου δηλαδή για την εκτέλεση δεν είναι υπεύθυνα ευρωπαϊκά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Δεν γίνεται δηλαδή άμεση διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Εκεί τότε εμεί έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία επίσης έχουν και αυτά θεσπίσει διαδικασίες ελέγχου της εκτέλεσης του προπολογισμού και επιθυμούμε να λάβουμε και τις δικές τους εμπειρίες. Όχι μόνο για λόγους ελέγχου των δικαιούχων, όχι για να δυσκολέψουμε τη ζωή κανενός, αλλά αντιθέτως για να εξηχνιάσουμε για ποιο λόγο σημειώθηκαν σφάλματα, για ποιο λόγο υπήρξαν καθυστερήσεις ενδεχομένως στην εκτέλεση του έργου του προγράμματος και για να μπορέσουμε να απαλείψουμε τα σφάλματα. Να μου επιτρέψετε να αρκεστώ σε αυτά σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να σηκώσετε απλώς και το χέρι και μπορείτε βεβαίως να τοποθετηθείτε και στην ε, μετρική σας γλώσσα, διότι έχουμε και τους γερμηνείς στη διάθεσή μας. Όταν κοίταξα το πρόγραμμα, σκέφτηκα δεν είναι δυνατόν να μιλούμε μόνο εμείς για δύο ώρες και να μην μιλήσει κανείς άλλος. Έχετε λοιπόν ευχαρίστω την δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις. Ορίστε, η Ινιές πρώτα Αγιάλα Σέντερ από την Ισπανία. Είμαι η σοσιαλίστρια εισηγήτρια για την Επιτροπή αυτή όσον αφορά την επερχόμενη απαλλαγή για τη χρήση 2017 ε, που ξεκίνησαμε τον Μάρτιο ε, του, και θα φτάσουμε τον Μάρτιο του 19. Οπότε και είχαμε εδώ επισήμω ε, το ελεγκτικό συνέδριο και βέβαια συνεργαζόμαστε τύπος όλο το χρόνο και με το Ελληνικό Συνεδρίο και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τέλος πάντων τώρα ήταν καθε αυτού η επίσημη διαδικασία για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε ό,τι χρειάζεται αυτό και μέσω των ε, ακροάσεων με τους ε, υποψηφίους επιτρόπους και να κάνουμε και την ετήσια έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Εκεί έχουμε δύο σημαντικά τμήματα. Πρώτα-πρώτα την ανάλυση, το νομικό έλεγχο για το τι έγινε κατά τη χρήση του 2017 και στη συνέχεια υπάρχει ο διάλογος, ε, η αντιπαράθεση ούτως υπήν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μοιάζει η διαδικασία με τη διαδικασία που ισχύει του εθνικού προπολογισμού. Αλλά επίση εμεί εδώ δουλεύουμε και στη βάση ενό πολιετού προπολογισμού. Ε, και μία από τις δουλειές είναι και η ανάκτηση ε, του τι έχει καταβληθεί αλλά και τι θα καταβληθεί κάποια χρόνια μετά. Και έχουμε και τη μέθοδο νη συν τρία. δηλαδή στο, σε κάποια οποιαδήποτε χρονιά θα έχουμε άλλα τρία χρόνια για την υλοποίηση των πολιτικών. Και στο τέλος, όταν η διαδικασία αυτή θα καταλήξει σε μια ισορροπία με για τον έλεγχο όλων των λογαριασμών, τότε έχουμε το πλήρες το οποίο ξεκαθαρίσει. Επομένω, για του χρόνου θα πρέπει να λάβουμε το ότι το 2017 ε, τελειώσαμε την πρώτη περίοδο προγραμματισμού, αρχίζει η επόμενη και έχουμε επομένως τώρα τους ελέγχους όσον αφορά τις ε, δαπάνες που αφορούν και την ε, κρίση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Επίσης, φέτος το 2018 ενώπιση 2019 παραλλήλως επεξεργαζόμαστε το νέο σχέδιο του πολιετούς προϋπολογισμού, αυτό που ονομάζουμε πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τον έλεγχο. Επότε, με τον έλεγχο που γίνεται, Θέλουμε στα πλαίσια της διαδικασίας της απαλλαγής να προβούμε σε παροχή συμβουλών και συστάσεων. Είμαστε ένα χρόνο πριν τις εκλογές και γι' αυτό και αυτή η απαλλαγή εξυπηρετεί κάτι σαν μέσον εξισορρόπησης ε, μεταξύ των εκλογών, της γνώμης του Κοινοβουλίου, ε, των όσων θα γίνουν το 9. Εξισορρόπηση, απολογισμός του ΣΥΠΗΝ και ταυτόχρονα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε αυτά που προβλέπονται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το Κοινοβούλιο και έχουμε επομένως κάποιον έλεγχο που πρέπει να είναι παραγωγικός. Έλεγχος ανά για διάφορα συστήματα τα οποία προβλέπονται και είναι συγκρίσιμα με κάποια συστήματα ελέγχου που ισχύουν και σε εθνικούς οργανισμούς και στα κράτη-μέλη. Έχουμε επίσης και τον έλεγχο επί των επιμέρους υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελέγχουμε τι αποτελέσματα παράγονται, τι είναι το πόσο είναι τέλο πάντων, το ποσοστό λάθος. Επομένως, έτσι γίνεται μια σειρά συνεδριάσεων όπως η σημερινή και καταλήγουμε στο τι γίνεται με το ποσοστό λάθους, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι γίνεται με τις πολιτικές που ασκούνται από κοινού με τα κρατημέλη, όπως οι πολιτικές συνοχής. Ε, τι γίνεται, ας πούμε, με κάποιες πολιτικές όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου. Τι γίνεται με την συγχρηματοδότηση γιατί υπάρχουν επιμέρους συστήματα σε κάθε οργανισμό, σε κάθε υπουργείο ε, και επίσης έχουμε κάποιες δικαιωτικές δομές διαφορετικές σε κάποια κρατημέλη όπως στην Ισπανία, όπου υπάρχει ένα σύστημα που προσυδειάζει σε κάθε διοικητική περιφέρεια και οι διοικητικές αρχές εκεί, οι διοικητικές περιφερειακές αρχές εκεί έχουν νομικές αρμοδιότητες Οπότε θέλουμε τα συστήματα να είναι όσο γίνεται πιο στεγανά, να επιδέχονται ε, έλεγχο, αξιολόγηση, να εμπνέουν αξιοπιστία. Όλα αυτά γίνανε και το 2017 για τις πολιτικές που ασκήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Οπότε ενίοτε χρειάζεται να αλλάξει ρότα ένας προϋπολογισμός, να διευρυνθεί, να προσαρμοστεί στις αυξανόμενες ανάγκες της συγκύριας. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μία φορά το χρόνο έχουμε την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και μας εξηγεί τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Και συνήθως έρχονται εδώ εκπρόσωποι του ελεγκτικού συνεδρίου και πολλές φορές ε, γίνεται η παρουσίαση με περιορισμένη σύνθεση της Επιτροπής οπότε και μαθαίνουμε πράγματα που δεν θα μαθαίναμε αλλιώ ότι συμβαίνουν. Και σας καλώ να παραστείτε στο βαθμό που μπορείτε σε αυτές τις παρουσίες του Ελληνικού Συνεδρίου και από πλευράς της δικής σας οπλικής γωνίας βοηθήστε μας επισημένοντας κάποια πράγματα που είναι χρήσιμα. Η πρόεδρος, ο κύριος Τσέλερ θέλει να συμπληρώσει κάτι. Ευχαριστώ, όχι ακριβώς συμπλήρωση. Ήθελα να ερωτήσω τους και τις συναδέλφους μας που είναι εδώ. Βρίσκω καλό ότι έχουμε κοντά μας κοινοβουλευτικούς συναδέλφους από χώρες που στοχεύουν στην ένταξη ή που συνδέονται μαζί μας μέσω της πολιτικής γειτονίας. Και στον τομέα αυτό ωραίουν σημαντικά κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Εδώ διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δίνονται χρήματα ιδίως στις κυβερνήσεις. Από όσο γνωρίζω, τα κονδύλια που δίνει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός σπάνια εμφανίζονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς των χωρών αυτών, αλλά τα διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις. Υπάρχει ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων, γίνεται ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων από τις κυβερνήσεις σχετικά με την ίσπραξη και διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και οι συνάδελφοί μας βουλευτές από τις διάφορες αυτές χώρες έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής αλλά και ελέγχου στην διαχείριση των χρημάτων αυτών. Αυτό για μας νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σαν βάση για μια μελλοντική καλύτερη συνεργασία. Η δική μου διαπίστωση είναι ότι συχνά στις χώρες αυτές και για θέματα περιφερικής ανάπτυξης. Η γνώση των κοινοβουλίων σχετικά με τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο που λειτουργεί είναι πολύ περιορισμένη. Η γνώση αυτή λοιπόν είναι πολύ περιορισμένη. Μάλιστα, θέσαμε μία ερώτηση. Υπάρχει κανείς εξημών που θα ήθελε να απαντήσει για λογαριασμό της χώρας του ή της Βουλής του. Δεν βλέπω μεγάλη προθυμία άχημα. Το ερώτημα λοιπόν, επαναλαμβάνει η Πρόεδρος, είναι εμπλέκεστε στη διαχείριση και έλεγχο της δαπάνης των κονδυλίων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων στις χώρες σας. Υπάρχει κάποιος από εσά που θα ήθελε να πει κάτι. Zahvaljujem. Ευχαριστώ. Από πλευράς Σερβικού Κοινοβουλίου να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χάραξη της δημοσιονομική πολιτικής για την επόμενη επταετία. και οι προοπτικές για την περίοδο 2021-2027 και για το ότι θα υπάρξει αύξηση προοικοδότηση για τα προγράμματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχω για τον οικονομικό και δημοσιονομικό έλεγχο κάτι να σας πω. Στην Σερβία έχουμε πολυεπίπεδο έλεγχο. Έχουμε εσωτερικούς ελέγχους για τους άμεσα και έμεσα δικαιούχους, έχουμε τους εσωτερικούς ελέγχους, την δημισιονομική επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης έχουμε την κεντρική υπηρεσία για τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και εκεί καθορίζεται η μεθοδολογία, γίνεται η κατάρτιση των αρμοδίων, αλλά έχουμε και εξωτερικό έλεγχο που γίνεται από την ε, Δημοκρατία Σερβίας, από το κράτος και συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως προαναφέρατε, η Επιτροπή σας, όπως και οι Εθνικές Επιτροπές Έλεγχου Προϋπολογισμού, έχει να επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο. Ο έλεγχος ε, κρατάει πολύ, δεν είναι κάτι πάρα πολύ δημοφιλές, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και είναι κάτι το οποίο επιτάσσει η εθνική νομοθεσία, αλλά και το εθνικό σύνταγμα. Μας είπατε ότι η Επιτροπή σας ασκεί έλεγχο για να επισημαθούν οι αντικανονικότητες για να διορθωθούν τα κακοσκήμενα αυτό αφορά και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και δις ετησίως υποβάλλονται σχετικές εκθέσεις από τους εισηγητές που αναλαμβάνουν τη σύνταξή τους. Έχω να σας ρωτήσω κάτι για αυτούς τους δείκτες επιδόσεων. Πολύ σημαντικό αυτό για τη λειτουργία και απόδοση του υπολογισμού. υπάρχουν κάποιες συστάσεις για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες για να αναδεχθούν, να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δείκτες ο καθένας στην χώρα του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και πέραν των ελεγκτικών μηχανισμών που μας αναφέρατε, σας αναφέρω επίση ότι έχουμε το λεγόμενο γραφείο προϋπολογισμού. Είμαστε η μόνη χώρα στα Δυτικά Βαλκανία, το μόνο κοινοβούλιο το οποίο έχει ε, μία πύλη στο διαδικτύο για αυτή την δουλειά. Είναι σημαντικά όλα αυτά για τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Αυτά ήθελα να σας πω, ξεκινώντας. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Αν καταλάβα καλά, είστε η κυρία Φιλιππόφσκη από τη Σερβία. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για το feedback που δώσατε. Έχετε άλλες παρατηρήσεις κάποιος άλλο. πολύ ευχαριστώ ε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Ε, ε, κάναμε και ταξίδι στην Σερβία ως Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού. σε κάθε περίπτωση θα τοποθετηθούμε και εμείς για την ορίμανση της πορείας προς την ένταξη μέσα στην οποία ε, τίθηκε το θέμα των δικτών. Βέβαια με τους δείκτες ασχολούνται πλήρωνε σε κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Πάντως εγώ έχω την πρόθεση να ζητήσω να εκφράσουμε κι εμείς συστάσεις, συστάσεις που θα προέρχονται και από τα εδάγματα προηγούμενων εντάξεων. Για παράδειγμα και χωρών όπως Ουγγαρία ή Πολωνία, με τις οποίες αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, ότι χρειαζόμαστε βιώσιμους μηχανισμούς ελέγχου και στις νεοεντασσόμενες χώρες, διότι αυτά που βλέπουμε είναι ότι οι χώρες κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να ενταχθούν και μόλις ενταχθούν χαλαρώνουν τις προσπάθειες, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Εάν θέλουμε να έχουμε βιωσιμότητα ως ένωση, πρέπει και οι ίδιες οι χώρες να καταβάλουν διαρκώς προσπάθειες και προσπάθειες επιτυχής και βλέπουμε από τις χώρες Βίσεγκραντ, Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, βλέπουμε από τη σύγκριση των χωρών αυτών ότι το ερώτημα ποιες προσπάθειες κάνει οι χώρες και πριν και μετά την ένταξη είναι σημαντική για την επιτυχία των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Την χειρότερη διαχείριση την κάνει η Ουγγαρία για την ώρα. Έχει σχέση με αυταρχικές κυβερνήσεις όταν έχετε απέναντί σας αυταρχικές κυβερνήσεις είναι δύσκολο ε, να, να επιτύχετε. Τα βλέπουμε αυτά από τις συγκρίσεις από, και από τους συγκριτικούς πίνακες που φτιάχνουμε και βλέπουμε ότι χρειάζεται διαρκής συνοδεία, δηλαδή να παραέχετε διαρκή συνοδεία και στις νέες χώρες. Δεν πρόκειται για ε, προσπάθεια ε, φήμωσης, πρόκειται αντίθετα για συνεργασία Χρειάζεται διαρκή έλεγχος και χρειάζεται και έλεγχος των διαδικασιών ελέγχου, αν είναι δυνατόν δηλαδή να βελτιωθούν. Τώρα, ο μηχανισμός έχει ακόμα πολλές αδυναμίες. Χρειάζεται λοιπόν να βελτιωθεί ο μηχανισμός της διεξαγωγής των ελέγχων, να βελτιωθεί πολύ και μέχρι ότου ενταχθούν οι χώρες σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρονικό αυτό διάστημα ώστε οι μηχανισμοί ελέγχου, οι μηχανισμοί της συνοδείας αυτής να βελτιωθούν σημαντικά. Δηλαδή εν μέρη μόνο είμαστε ικανοποιημένες και ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Βλέπετε και την κατάσταση στη Ρουμανία με τον μηχανισμό συνεργασίας και επαλήθευσης που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Άλλοι επιθυμούν να τοποθετηθούν από τη δική σας πλευρά. Θάρρο, θάρρο. Δεν ε, δαγκώνουμε. Με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε τις απόψει σα. Θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Σμιτ για την απαλλαγή του, Ευρω... του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Ε, προσοχή, καμιά φορά δαγκώνουμε κιόλας. Υπενθυμίζω πώς έχει δημιουργηθεί ο κοινοβουλευτισμός τον 12ο αιώνα υπήρχε ένας βασιλέας ο οποίος ήταν υπερβολικά γενναιόδωρος στις δαπάνες, χρειάστηκε να αυξήσει την φορολογία, οι βαρόνοι δεν συμφώνησαν, πήγαν λοιπόν και του είπαν έλα εδώ, τον πιάσαν από τα αυτιά ή τον δάγκωσαν, δεν ξέρω τι ακριβώς έκαναν, εν πάση περιπτώσει δεν τον άφησαν να συνεχίσει να είναι το ίδιο αλαφρόμυαλος. Το ίδιο λοιπόν και εμεί εδώ οι κοινοβουλευτικοί οφείλουμε να παίξουμε το ρόλο των βαρώνων του 12ου αιώνα. Καμιά φορά δεν μας συμπαθούν τόσο πολύ, όταν δηλαδή κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δηλαδή πάμε και ελέγχουμε όλους εκείνους που δαπανούν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και εξετάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά το τι κάνουν, διότι αυτό είναι το καθήκον μας. Όπως είπε ήδη η Πρόεδρός μας, πάντοτε τους βρίσκουμε αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Ακούσαμε ήδη από τους συναδέλφους που μίλησαν προηγουμένως το πώς διεξάγεται ο έλεγχος των δημοσιονομικών. Εγώ εισηγήτρια είμαι για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ίσως σας φανεί λίγο ασυνήθιστο, διότι ε, αυτοελέγχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελέγχει δηλαδή το ίδιο τις δαπάνες του και χορηγεί απαλλαγή στον εαυτό του. Ακούσαμε όμως από τους συναδέλφους μας ότι ο χρόνος για την χορήγηση της απαλλαγής αρχίζει με την δημοσίευση της ετήσιας εκθέσεως του Ελεκτικού Συνεδρίου, αρχές Νοεμβρίου, που αποτελεί και τη βάση για την περαιτέρω Και μετά τοποθετούνται οι Γενικέ Διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι και τον ίδιο τον Επίτροπο και γραπτό και προφορικό. Μετά γίνονται τροπολογίε. Η δε τελική έκθεση καταλήγει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό γίνεται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτου. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τότε. Η απαλλαγή, αυτά για τον κανονικό προπολογισμό τη Ένωση. Ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δεν προβλέπει συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο προβλέπει συνεργασία με τον πολύ ισχυρό Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κλάους Βέλε, ο οποίος τον Νοέμβριο μας δίνει έκθεση για το follow-up των εκθέσεων που έχουν ψηφιστεί την προηγούμενη χρονιά. Μετά συντάσσεται κατάλογος ερωτήσεων από όποιον ενδιαφέρει και τέλος Ιανουαρίου γίνεται σχετική ακρόαση για τις ερωτήσεις που έχουν υποβάλει οι ευρωβουλευτές. Το υπόλοιπο κινείται στις ίδιες γραμμές όπως η απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τον Νοέμβριο, τον του ενός έτους μέχρι τον Απρίλιο του επομένου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως είπα είμαι η συγγήτρια για τον έλεγχο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 2017. Εδώ οι δαπάνε του Κοινοβουλίου ανήλθαν στο 1,75 δισεκατομμύριο ευρώ. Χρήματα έχουν δοθεί για, ε, ε, για ε, πολιτικές εργασίες, έχουν δοθεί για κτίρια και πάνω από 50% για δαπάνες προσωπικού. Πρόκειται κατά βάση για διοικητικό προϋπολογισμό, αντίθετα με τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό που ε, δαπανά τα χρήματά του, τα κονδύλια του για έρευνα, για παράδειγμα, για εκτελεστικά προγράμματα κλπ. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα και εμένα και τις ε, συναδέλφους μου κάθε χρόνο, που εμφανίζονται ξανά και ξανά κάθε χρόνο και όπου δεν φαίνεται να λύνονται τόσο γρήγορα, όπως για παράδειγμα αφενός το συνταξιοδοτικό ταμείο των πρώην Ευρωβουλευτών, το οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχει και το οποίο κάθε χρόνο επανέρχεται ως πρόβλημα, διότι είναι πάντοτε στο μείον. Έχουμε προεδρείο, του οποίου ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, υπάρχουν οι 14 αντιπρόεδροι και 5 κοσμήτορες. Εκεί διεξάγονται δύο συνεδριάσεις τον μήνα και στο Προεδρείο αυτό λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι μέχρι ότου εφαρμοστούν οι αποφάσεις, εμείς οι Ευρωβουλευτές δεν γνωρίζουμε τι έχει συζητηθεί στη συνεδριάση του Προεδρείου, πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί δυνάμεων, ποιος λαμβάνει τις πρωτοβουλίες για τις διάφορες αποφάσεις. Ένα απλό παράδειγμα. Το Κοινοβούλιο έχει ένα στολίσκο οχημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμός αναλαμβάνει, ας το πω διαφορετικά, έχουμε λοιπόν το στόλο των οχημάτων. Είναι πολύ μεγάλος. Έχουμε τώρα προσλάβει εμείς οι ίδιοι τους οδηγούς. Δεν είναι πλέον outsourcing, δεν ανατίθεται σε εξωτερική εταιρεία και αυτό για λόγους ασφαλείας των ευρωβουλευτών. Τώρα όμως δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει παραπέρα με τον στόλο των οχημάτων. Όλοι έχουμε τους στόχους του περιβάλλοντος, του κλίματος κλπ. Έχουμε περάσει σε ηλεκτροκίνηση ή σε υβριδικά οχήματα σε ένα μεγάλο βαθμό του στόλου, αλλά δεν ξέρουμε πού θα πάει. Έχουμε σκεφτεί να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα αυτά και ενδεχομένω συνθετικά καύσιμα στο μέλλον, δεν ξέρουμε. Όμως ποιε θα είναι οι μελλοντικέ εξελίξει. Πράγματα τα οποία οι δύο ευρωβουλευτέ, αν ερωτήσουν, δεν λαμβάνουν απαντήσει. Εάν όμω είναι κανεί εισηγητή, όπω είμαι εγώ τώρα εισηγήτρια, δηλαδή, εάν θέσω ερωτήσει σε οποιαδήποτε διεύθυνση, αμέσω λαμβάνω απαντήσει και απαντήσει σε βάθο. Εγώ διακρίνω και μια αυθαιρεσία βέβαια εδώ στη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Δεν ακολουθούν όλοι τους ίδιους κανόνες, δηλαδή βλέπεις ότι ορισμένα πράγματα χρειάζεται μόνο μια υπογραφή, αλλού αρκεί το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου. Όλα αυτά είναι αδιαφανή, εάν κανείς δεν τα εξετάσει από πιο κοντά. Και βεβαίω τίθεται πάντοτε και το ερώτημα τι γίνεται στις διοικητικές μονάδες του Κοινοβουλίου και τι θα πρέπει να συμβεί και στα γραφεία των Ευρωβουλευτών. Ένα από τα πιο δαπανηρά προβλήματα, θα το ακούσατε ίσως ήδη, συχνά μιλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτό το τσίρκο, το περιπλανόμενο τσίρκο, διότι μια φορά το μήνα, μια εβδομάδα, την περνούμε στο Στρασβούργο, όπου είναι η μία από τις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εκεί ταξιδεύουν λοιπόν ευρωβουλευτές, ε, βοηθοί των ευρωβουλευτών, άλλοι συνεργάτες, που φτάνει σε τριψήφιο ποσό τον εξαψήφιο δηλαδή ποσό τον χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως περιττή αυτή η μετακίνηση. Άλλοι υπάρχουν βεβαίως που το ζητούν. Υπάρχει από παλαιά σχετική συμφωνία, Ποιος είδε τι γίνεται και με το Brexit και πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει μια συνθήκη, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι και αυτό το εγχείρημα. Οι διοικητικέ διαδικασίες αμφισβητούνται συχνά, καθώς και το κόστος τους. Οφείλει να λαμβάνει κανείς υπόψη βέβαια ότι μιλεί για μια τεράστια διοικητική μηχανή, επίσης με μια μεγάλη ακίνητη περιουσία. Το 78% όλων των κτηρίων όπου είναι του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ιδιοκτησία του. Για παράδειγμα, τα γραφεία πληροφοριών, συνδέσεων σε διάφορες χώρες μέλη. Επίσης, τα κτίρια εδώ στο Βέλγιο, τα κτίρια του Στρασβούργου και βεβαίως και κάποια κτίρια στο Λουξεμβούργο. Και το ερώτημα βέβαια που τίθεται εν τέλει είναι πώς γίνεται η διαχείριση των κτίριων αυτών, διότι αφενός είναι μια μεγάλη περιουσία, από την άλλη μεριά βέβαια έχει και κόστος η συντήρηση των κτηρίων αυτών και ούτω καθεξής. Η απαλλαγή λοιπόν, η χορήγηση απαλλαγή για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όταν ως εισηγήτρια ασχοληθεί κανείς με αυτήν την διοίκηση και βλέπει τι γίνεται και στα πλαίσια και ε, παράπλευρα ε, με αυτήν την κοινοβουλευτική εργασία βλέπει και πόσα ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα γίνονται ωστόσο και διαπιστώνει κανείς ότι και σε ορισμένε διευθύνσει υπάρχουν κάποιες προτιμήσεις υπέρ κάποιων χωρών μελών. Για παράδειγμα, για το προσωπικό ασφαλείας βλέπουμε περισσότερους Βέλγους, Γάλλους και Ρουμάνους. 400 από 520 δηλαδή υπαλλήλου της ασφαλείας είναι από αυτές τις χώρε. Μια λοιπόν ελίπουσα γεωγραφική κατανομή. Έχει διάφορους λόγους ε, αυτό το πράγμα. Αυτό που εξετάζουμε εμείς και μπορώ να το πω ότι το Προεδρείο θα συμφωνήσει η διοίκηση του Κοινοβουλίου εργάζεται καλά. Υπάρχουν βέβαια αδυναμίες, μου λένε καμιά φορά είσαι κακιά διότι κοιτάς τι δεν λειτουργεί σωστά. σου κοιτάζω και αυτό. Είναι σωστό να θέτει κανείς τον δάκτυλο επί των τύπων των ήλων, διότι δεν είναι δυνατόν εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού, να ελέγχουμε τον προϋπολισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά εδώ στο δικό μας προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να κλείνουμε το ένα μάτι. Έχω δει λοιπόν κάποια γκρίζα ή μαύρα σημεία τα οποία θα τα θέσω στην έκθεσή μου. Πάντως στο σύνολό τη η διοίκηση του Κοινοβουλίου εργάζεται καλά. Βλέπετε ότι οι διερμηνείς μας απεργούν παρόλο που εργάζονται. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ανεξαρτήτως του τμήματος. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα τώρα μετά από όλες αυτές τις επιθέσεις που έγιναν και εδώ στις Βρυξέλλες είτε στην υπηρεσία των οδηγών είτε στην υπηρεσία των μεταφράσεων. Γίνεται πράγματι ε, σπουδαία δουλειά και όπου υπάρχουν αδυναμίες εμείς τις εντοπίζουμε και ελπίζω ότι με κοινή προσπάθεια θα τις διορθώσουμε. Yeah, σας ευχαριστώ. Αν έχετε ερωτήσεις, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι παρατηρήσεις. Βλέπω από τις λεπτομέρειες που ακούσαμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση χορήγηση απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Ερώτηση προς τις και τους συναδέλφους. Τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί το θέμα για τη δεύτερη αυτή συνάντησή μας επίδοση και ορατότητα ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμεθοριακή συνεργασία. Επειδή είμαι μέλος και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης όπου τα διορθωτικά ταμεία σε ό,τι αφορά ε, την οθετική τους βάση εκεί εγκρίνονται, είναι δικό μας αίτημα στην παρούσα περίοδο στήριξης να τονίσουμε ιδιαίτερα την διαμεθοριακή συνεργασία όχι μόνο μεταξύ περιφερειών εντός των χωρών μελών της Ένωσης, αλλά διαμεθοριακή συνεργασία και προς γειτονικέ χώρες, γειτονικέ τρίτες χώρες και να ανοίξουμε τα μέσα και τα όργανα που διαθέτουμε. Και στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία αυτή. Και όπου είναι δυνατόν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου διαπιστώνω ότι υπάρχουν ακόμα φραγμοί λόγω των διαφορετικών εθνικών νομοθετικών συστημάτων. Δημιουργήθηκε ιδιαίτερο νομοθέτημα για την συνεργασία των περιφερειών που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον ωραίο κάπως μπαρόκ τίτλο Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαμεθοριακή συνεργασία. Αν όμως δω τον χάρτη εν τέλει, έχουμε 60 τέτοιες συνεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η διαμεθοριακή συνεργασία προς γειτονικέ χώρες είναι ακόμα πάρα πολύ περιορισμένη. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια συνεργασία μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας, που είναι γειτονική τρίτη χώρα. Δεν βλέπω εκτός από αυτό και πάρα πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Το θέμα αυτό συζητείται παροιμήν, με ύψιλον δηλαδή. Και για τον κόσμο, για τους ανθρώπους είναι ενδιαφέρον, όχι μόναχα δηλαδή η ελευθερή κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκεί όπου υπάρχουν περιφέρειες που δεν έχουν και μεγάλες διαφορές εκατέρωθεν των συνόρων, ούτε οικονομικές, ούτε πολιτικές, ούτε πολιτιστικές. Και εκεί υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν διάφορα ταμεία και διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και μπορεί να, να ζητηθεί και η συνδρομή τους και για τη διαμεθοριακή συνεργασία. Έχουμε νέες προτάσεις κανονισμών Υπάρχει και νέος κανονισμός που προβλέπει εκεί όπου υπάρχουν ακόμα φραγμοί στην διαμεθοριακή συνεργασία, αυτοί οι φραγμοί να μειωθούν έτσι περαιτέρω. Εάν εγκριθεί το σχέδιο κανονισμού που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει νομοθεσία της Ένωσης, αλλά και μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων Interreg της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Συνεργασίας όπου συνεργάζονται πανεπιστήμια, άλλοι φορείς και μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Στοχεύουμε σε διευκόλυνση αυτών των συνεργασιών. Εδώ θα χρειαστεί αναγκαία η συνεργασία μαζί σας. Η εργασία αρχίζει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα χρειαστεί ανταλλαγή απόψεων και μαζί σας και αν έχετε τη σχετική προθυμία και διάθεση να ενισχύσετε τη διαμεθοριακή αυτή συνεργασία και να αναζητήσετε νέους δρόμους μαζί μας. Αυτό θα είναι βέβαια ιδιαίτερα χρήσιμο για την συνεργασία και για τη συμβίωση τελικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανεξαρτήτως διαπραγματεύσεων για ένταξη, τις οποίες χειρίζονται οι κυβερνήσεις, παρόλα αυτά μπορεί να ενισχυθεί η εργασία αυτή, η διαμεθοριακή δηλαδή συνεργασία, πριν ακόμα από την ολοκλήρωση της ένταξης. Εν προκειμένου, επισημαίνω ότι για την εξωτερική πολιτική θα υπάρξει γενικός κανονισμός, στον οποίο θα περιληφθούν όλα τα σχετικά μέσα για την αναπτυξιακή συνεργασία, για την υποστήριξη των, ε, της, της πορείας της, για την ένταξη, πολιτική γειτονία, όλα αυτά δηλαδή θα μπουν κάτω από μια ομπρέλα, σε ένα ενίο νομοθέτημα, με σαν ανατομέα πολιτικής. Αλλά μετά θα πρέπει κανείς να αναζητήσει που βρίσκονται οι προκλήσεις, προκλήσεις όπως τώρα ας πούμε έχουν προκύψει από το μεταναστευτικό, ώστε να μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα και οι θεσμοί, η Κομισιόν είναι προκειμένου. Άλλωστε λέμε συχνά όποιος ε, ξυπνάει νωρίς και πιάνει νωρίς δουλειά έχει και μεγαλύτερη επιτυχία. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν για τους τομείς αυτούς πολιτικής. Γι' αυτό εν τέλει το ερώτημα που επιθυμώ να σας θέσω είναι αν μπορεί να ενισχυθεί αυτή η διαμεθορική συνεργασία κατά τη γνώμη σας. Η Πρόεδρος, να μεταφέρουμε την ερώτηση αυτή στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης, γιατί έχουμε τώρα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τη συνεργασία στα Αυτό, στα Δυτικά Βαρκάνια μάλλον. Αυτά γίνει μετά. Τώρα έχουμε τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο δεύτερο μέρος ακροάσεως θα εμβαθύνουμε στη συνερώτηση που κάνατε. Τώρα ο κύριος Κον για τις απαλλαγές των προϋπολογικών. Ευχαριστώ πολύ. Απευθύνω χαιρετισμό στην αλβανική γλώσσα κάποιες λέξεις καταλαβαίνω από αλβανικά και από σερβικά, ε, γι' αυτό τις χρησιμοποίησα. Λέγομαι Κον, είμαι από το Άχεν στην Γερμανία, Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Είμαι και μέλος στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Δεν είχα τη χαρά να βρεθώ στην Αλβανία ως τώρα, αλλά με την πρόεδρό μα και με την κυρία Τζαβάλοβα ε, πήγαμε στην ε, Σερβία και στην Κροατία την προηγούμενη χρονιά και έχω έτσι μια πρώτη εικόνα από τις χώρες σας. Χαίρομαι που είστε παρούσες και παρόντες και σας κάνουμε ένα είδος εντατικό φροντιστήριο για ευρωπαϊκά θέματα. Και πραγματικά ε, σας βγάζω το καπέλο που βλέπω να παρακολουθείτε ε, τόσο προσεκτικά, διότι βέβαια δεν είστε τόσο γνώστες του θέματος όσο εμείς. Έρχομαι στο θέμα, ε, το δικό μου τώρα, είμαι εισηγητής για το έτος 2017 για την απαλλαγή των λοιπών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δηλαδή όλων των θεσμικών οργάνων με εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπου όπως ακούσατε προηγουμένως είναι ξεχωριστές οι απαλλαγές. Άρα δηλαδή μιλούμε για την Επιτροπή Περιφερειών, που είναι το θεσμικό κοινό όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δήμαρχοι, περιφερειάρχες και το καθεξής, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, κοινωνικοί εταίροι κλπ. Το Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαίος, ε, Ευρωπαϊ, Εντεταλμένος Προστασία των ε, Προσωπικών Δεδομένων, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα άλλα λοιπόν, τα λοιπά θεσμικά όργανα, είναι υπόλογα κάθε χρόνο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς εξετάζουμε τις δαπάνες τους πάρα πολύ προσεκτικά. Στο μέγα μέρος είναι διοικητικές οι δαπάνες αυτές. έρχονται στο σύνολο του 6% του συνολικού ευρωπαϊκού προπολογισμού, του συνολικού ενωσιακού προπολογισμού. Δηλαδή πολύ περιορισμένο ποσοστό. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό ε, να αποδείξουν τα θεσμικά αυτά όργανα ότι δαπανούν νομότυπα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που λαμβάνουν. Διότι η σωστή διαχείριση του προπολισμού είναι αναγκαία απέναντι στον πολίτη. Διότι ο πολίτη ε, πρέπει να έχει την αίσθηση ότι σωστά χρησιμοποιούμε τα χρήματά του, είναι φορολογούμενο. Μέγα μέρο των προπολογισμών βέβαια δαπανώνται για δαπάνε προσωπικού, υπάρχουν μετά δαπάνε ίδρυση κτηρίων, μετάφραση, ε, άλλε λογιστικέ δαπάνε κ.ο.κ. Και εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι τελικά είμαστε όλοι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχει κανείς τη δυνατότητα να δει τι ακριβώς, ε, ποια είναι τα πράγματα εκείνα που συναποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι για ποια πράγματα. Ως εισηγητής λοιπόν έρχεται κανείς σε επαφή με εκπροσώπους όλων αυτών των θεσμικών οργάνων, ε, ανταλλάσσει απόψεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια χαίρει μεγάλη εκτιμήσεω, διότι εμεί είμαστε εκείνοι οι οποίοι εν τέλει θα δώσουμε τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα να διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια για να εκτελέσουν τα καθήκοντά του. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια είμαστε και σύμμαχο των θεσμικών οργανών. για την ε, υπεράσπιση των προϋπολογισμών τους απέναντι στις χώρες μέλη, διότι συχνά οι χώρες μέλη έχουν το ενδιαφέρον να μειώσουν όσο το δυνατόν τις δαπάνες της Ένωσης και επομένως την συνεισφορά τους στο Ταμείο της Ένωσης. Εγώ θεωρώ πάντως ότι κανείς δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από το τίποτα. Δηλαδή άμα δεν θες να δαπανίσεις τίποτα, δεν θα λάβεις και τίποτα. Δεν μπορεί να αναμένει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει χωρίς τα αναγκαία κονδύλια. Επομένω, και τα θεσμικά όργανα που προανέφερα θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή του τα απαραίτητα κονδύλια για να εκτελούν τα καθήκοντά του. Φροντίζουμε και προσέχουμε ωστόσο να γίνεται σωστά η διαχείριση των κονδυλίων, να εκμεταλλεύονται κάθε δυνατότητα εξοικονόμηση, Για παράδειγμα, συστεγάζονται σε κτίρια ορισμένα, ορισμένοι από τους θεσμούς αυτούς. Έχουν γίνει και συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κοινή χρήση των μεταφραστικών υπηρεσιών. Ε, κάνουμε λοιπόν προσπάθεια εξοικονόμησης και αποτελεσματικής, αποδοτικής δαπάνης των χρημάτων. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το καθήκον να επισημαίνουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν θεσμικά όργανα όπου, για παράδειγμα, απασχολούνται ασκούμενοι ε, χωρίς αμοιβή ή όταν δεν είναι σωστή η κατανομή αναφύλω. Υπάρχουν ε, άλλα τέτοια προβλήματα. Για παράδειγμα, η γεωγραφική κατανομή, αναεθνικότητα, όπου καμιά φορά δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες. Εμείς τότε είμαστε εκείνοι οι οποίοι λέμε, οι ευρωβουλευτές δηλαδή, α, προσοχή, εδώ υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να διορθωθεί. Η μοναδική εξαίρεση σε αυτή την καλή συνεργασία είναι το Συμβούλιο το οποίο έω τώρα, το Συμβούλιο Υπουργών δηλαδή, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό έω τώρα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω και εδώ έχουμε αρχίσει να βελτιώνουμε την κατάσταση. Η πρόεδρό μα διεξάγει συζητήσει μαζί με του συναδέλφου ε, Βέλγου ευρωβουλευτέ, ώστε να επιτύχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο των Υπουργών, ώστε στο μέλλον και το Συμβούλιο Υπουργών να λαμβάνει χορήγηση απαλλαγής για τον προπολογισμό του από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις για τα όσα μόλις σας εξήγησα και σας ενθαρρύνω να θέσετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Συνεχίζομαι με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Ο κύριος Σάρβαμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέγομαι Πέτρη Σάβαρμα. Είμαι πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών και συντονιστής ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, σε αυτή την Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού. που φυσικά είναι η καρδιά του κυρουβλίου. Αν ε, δούμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για το αν ε, πράττουν βάση νόμου και αν εκτελούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση. Χωρίς να επαναλάβω πολλά που έχουν υποθεί και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Χαίρομαι που σας βλέπω σε όλους σε αυτή την επιτροπή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, χωρίς να επαναλάβω τώρα, θέλω να πω κάτι που αφορά την διαδικασία απαλλαγής εν γέννη. Είναι μια λεπτομερής και ενορχιστρωμένη διαδικασία. Αυτή η Επιτροπή υλοποιεί ακροάσεις των ε, φορέων που είναι υπό εξέταση και τους ε, ασκούμε μεγάλη κριτική και επικοδομητική αλλά και αρνητική σε ορισμένες περιπτώσεις. Το αν θα χορηγήσουμε την απαλλαγή ή θα την αναβάλουμε είναι πάντοτε μία απόφαση κατόπιν ορίμου σκέψεως. Και πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι αν δεν χορηγήσουμε την απαλλαγή αυτό αποτελεί ένα πολύ ισχυρό πολιτικό εργαλείο για τη διόρθωση των παρατυπιών και των προβλημάτων στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Αν δεν είναι αν δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι λογαριασμοί, θα πρέπει ο εν να ακολουθήσει τις συστάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού πριν να ξαναζητήσει απαλλαγή. Και η χορήγηση της απαλλαγής δίνει ένα θετικό μήνυμα της αποτελεσματικής εφαρμογής και δαπάνης των χρημάτων των φορολογουμένων. Όπως είπε και ο κύριος Κον, συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό εργαλείο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής και εξετάζει τις παρατυπίες στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού καθώς και τα μέτρα πρόληψης και έρευνας τέτοιων περιπτώσεων. Τώρα θα σας πω δύο λόγια για τους οργανισμούς, τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το θέμα της συζήτησής μας. Εγώ δύο φορές ήμουν σκιώδης για το ΕΛΚ, για τους οργανισμούς και ήμουν συζητητής του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή για το 2012 και τώρα πάλι εμείς για το έτος 2017. Τι είναι οι οργανισμοί για να ξεκινήσουμε. Βοηθούν την Ευρώπη να γίνει ένα καλύτερο μέρος. Μπορεί να το πει κάποιος έτσι πολύ απλά. Όμως, κάνουν πολλά. Οι οργανισμοί έχουν συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υλοποιούν τεχνικά και επιστημονικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν πολιτικές και να λάβουν αποφάσεις. Βρίσκονται σε όλη την Ήπειρο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργάζονται επί θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών, των 500 εκατομμυρίων πολιτών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο παρέχοντας ε, στα θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη ειδική γνώση σε τομείς ε, που είναι ποικίλοι. Κυμαίνονται από ε, το θέμα της διατροφικής ασφάλειας, από την έφησα μέχρι τα φάρμακα που παίρνουμε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, το σχάρι, μέχρι τα χημικά με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών, η CHA, και έχουν έδρα σε διαφορετικές πρωτεύουσες των κρατών μελών ή σε πόλεις. Και Φυσικά ε, έχουμε και το θέμα των μεταφορών, την ποιότητα των συνδικών εργασίων μας, ε, το περιβάλλοντος, 32 ε, οργανισμούς έχουμε συνολικά. Και το ουσιαστικό σκέλος ε, του ελέγχου και της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού είναι να εξετάζουμε και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Αυτοί οι αυτόνομοι οργανισμοί έχουν πολιτική εντολή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ανεξάρτητα και να εφαρμόζουν τον προπολογισμό της Ένωσης στον τομέα πολιτικής τους. Απολυθούν ουσιαστικό τμήμα της πολιτικής δομής της Ένωσης και οι δράσεις τους πρέπει να ακολουθούν φυσικά τους κανόνες και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δουλειά του Κοινοβουλίου εδώ ως αρμόδια αρχή για την απαλλαγή είναι να ελέγχει ότι όλες αυτές οι πτυχές λαμβάνονται υπόψη στο έργο των οργανισμών. Έτσι λοιπόν έχουμε ακροάσεις ε, μαζί τους, έχουμε επισκέψεις επιτόπου στους οργανισμούς και έχουμε ε, ερωτηματολόγια λεπτομερή που κάθε χρόνο πρέπει να απαντούν. Και επικοδομητικές συζητήσεις και φυσικά συνεδριάσεις με το προσωπικό. Τους συναντάμε, συνεχώς έρχονται εδώ. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή Ελέγχου του Προεπιλογισμού με το πέρασμα των ετών έχει υλοποιήσει κάποιες συστάσεις για διάφορα ζητήματα. Τυπικά, χαρακτηριστικά, μπορεί να, μπορεί να πρόκειται για αδυναμίες στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν τους οργανισμούς ή αδυναμίες Ω προς το θέμα του ετήσιου χαρακτήρα του προπολογισμού, των μεταφορών, των κονδυλίων ή των ακυρώσεων. Εξετάζουμε την πολιτική που έχουν για το προσωπικό, το θέμα της διαφάνειας, τους ιδρικούς ελέγχους κτλ. Και ο στόχος της δουλειάς μας δεν είναι να μικροδιαχειριζόμαστε την καθημερινή δουλειά των οργανισμών, αλλά παρακολουθούμε την Επιτροπή του Προπολογισμού και να δίνουμε πολιτική καθοδήγηση για την εκτέλεση των καθηκόντων και των εντολών των οργανισμών. Η Επιτροπή μας δίνει μεγάλη έμφαση στις επιδόσεις παρά να εξετάζει απλά τα νούμερα και τις δαπάνες. Γιατί θέλουμε να δούμε αντίκτυπο και αποτελέσματα. Αυτά θέλουμε να επιδεχάνονται με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και των χρημάτων των φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε κάτι ακόμα, έχουμε τα joint undertakings, η κυρία Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και πάλι, λέει η κυρία Τιμπάλοβα. Προέρχομαι από τη Δημοκρατία, ένα από τα κράτη-μέλη που εντάχθηκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Εξακολουθεί να είναι πρόσφατη η εμπειρία μα για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία να ανταλλάξουμε μαζί σα. Μεγάλη πείρα. Είμαι και εγώ αντιπρόεδρο αυτή τη επιτροπή και όπως σας είπα είναι μια αρκετά δύσκολη επιτροπή. Όμως αυτό που μου αρέσει είναι αυτή η οριζόντια ε, άποψη αυτών των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί και τι συστήνουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό. Θεωρώ αυτό το training, αυτή την κατάρτιση πολύ καλό για όλους μας ε, και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. πρέπει να το κάνουμε και για μας, γιατί χαίρομαι προσωπικά που ακούω όλες αυτές τις διαδικασίες απαλλαγής, πώς οργανάζονται και πώς το βλέπουν οι διάφοροι συγητές. Ήμουν πολύ τυχερή που ήμουν συγητρία για την ε, απαλλαγή. Είναι ε, ήταν αυτό το δεύτερο χρόνο της ε, πολιτικής μου πείρας. Έτσι λοιπόν είχα μια καλή επισκόπηση των πάντων και της συνεργασίας εδώ. Και πάντοτε ε, παρέμεινα σκιώδης ε, για την απαλλαγή της Κομισιόν και για τον κοινοπραξιών και φέτος είμαι συγγήτρια για τις κοινοπραξίες. Ακούσατε λοιπόν πολλά για τη διαδικασία της απαλλαγής, τώρα θα αναφέρω κάτι για τις κοινοπραξίες. Τι, σε τι συνίσταται και είναι πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε γιατί συστάθηκαν οι κοινοπραξίες και πώς λειτουργούν. Ορίζονται από το άρθρο 187 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόκειται για συγκεκριμένες δομές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση της ε, έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης ε, και των ε, προγραμμάτων επίδειξης. Τα μέλη των κυριοπρασιών είναι τυπικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιες βιομηχανικές ενώσεις, καθώς και άλλοι εταίροι που είναι ενεργοί στην έρευνα και στην ανάπτυξη κοινοπραξίες έχουν το δικό τους θεματολόγιο για την έρευνα και ζητούν χρηματοδότηση βάση ανοιχτών ε, προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Δηλαδή έχουν τους δικαιούχους τους δικούς τους, ε, ξεκινά διαγωνισμός και παραχεται χρηματοδότηση. Κάποια τυπικά χαρακτηριστικά και θα ξεκινήσω με την ε, μεγάλη και θα μιλήσω αργότερα για τα χρήματα είναι το Fusion for Energy ή μπορείτε να το ξέρετε ως ίτερ. Είναι η κοινοπραξία που είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία και το συντονισμό για το σχεδιασμό, την έρευνα, την ανάπτυξη και την ε, κατασκευή των ε, μεγαλύτερων ε, ουσιαστικά μερών που χρειάζεται για την κατασκευή του ίτερ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει μέχρι το 50% του κόστους και εδρεύει στην Γαλλία. Το δεύτερη τυπική κοινοπραξία είναι ο νέος ευρωπαϊκός ε, ουρανός ε, και σχετική έρευνα λέγεται ΣΕΖΑΡ και αναπτύσσει τη νέα γενιά των ε, νέων συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας κυκλοφορίας. Μετά έχουμε άλλα έξι ειδικά είδη κοινοπραξιών, κοινέ κοινοπραξίε, κοινέ τεχνολογικέ πρωτοβουλίε έχουν συσταθεί για να εφαρμόσουν ένα μέρο του θεματολογίου στην έρευνα. Λέγονται JTIs. Και κυρίως προκύπτουν από τη δουλειά κάποιων πλατφόρμων. Έχουμε περνούν το χάρη καινοτόμα φάρμακα, μπορείτε να φανταστείτε. Ε, μιλάμε για φάρμακα, θεραπείες, αντιβιωτικά, παραδείγματος χάρη, ε, υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου. Ε, για να έχουμε πράσινες και αποτελεσματικές τεχνολογίες, τις μεταφορές καθαρό ουρανό, αναπτύσσει ε, κάποια πιο ελαφρά ε, αεροπλάνα με χαμηλότερες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα και μετά έχουμε τις ε, βιολογικές βιομηχανίες, έχουμε ε, τα ηλεκτρονικά ε, συστήματα για την πρόθεση των ηλεκτρονικών ικανοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τελευταία είναι το Shift to Rail ε, που αναπτύσσει καλύτερε υποδομέ, σιδηροδρομικέ ε, για να μειωθεί το κόστο και να βελτιωθούν οι ικανότητε και η αξιοπιστία των τρένων. Αυτέ είναι οι οκτώ κοινέ κοινοπραξίες κοινοπραξίε, με που πρέπει φυσικά να ελέγχονται από την Επιτροπή μα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση με τον συνολικό προπολογισμό των κοινοπραξιών. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, όχι ένα έτο, αλλά σύμφωνα με το σημερινό πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ε, η επταετή προγραμματική περίοδο που θα ολοκληρωθεί το 2020. Όλο το PDP είναι 1,87 ε, δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε 10 δισεκατομμύρια για τις κοινοπραξίες, δηλαδή 0,9% του συνολικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για να έχετε μία ιδέα για τον προϋπολογισμό των κοινοπραξιών. Η μεγαλύτερη, όπως σας είπα, είναι το Fusion for Energy, το ITER, και έχουμε για τον προπολογισμό για την επταετή περίοδο είναι 3 δισεκατομμύρια και αποτελεί το 0,27% όλου του προπολογισμού του PDP. Αυτό είναι για να έχετε μια ιδέα για το μέγεθος και για τα χρήματα. Τώρα, ποιες είναι οι κυρίες προκλήσεις που έχουμε με τη διαδικασία απαλλαγής των κοινοπραξιών. Θα σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα των τελευταίων διαδικασιών απαλλαγής που είχαμε για τις κοινοπραξίες και στη συνέχεια θα ήθελα να κλείσω με κάποια γενικά σχόλια για τι κοινοπραξίε και την ορθή διαχείριση. Καταρχήν, ένα από τα προβλήματα στη διαδικασία απαλλαγή για τι κοινοπραξίε είναι ότι δεν υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ των προγραμμάτων πλαίσιο που επικαλύπτονται ε, από δύο και παραπάνω έτη. Οι, εφαρμο... πληροφορίες δηλαδή σχετικά με την εφαρμογή και οι δείκτε δεν διασφαλίζουν την πραγματική αξιολόγηση των επιδόσεων εγκαίρω, γιατί υπάρχει αυτή η επικάλυψη. Στη συνέχεια, ένα μεγάλο πρόβλημα σε κάποιε κοινοπραξίε είναι ε, το θέμα των προμηθειών, ε, κυρίως όταν έχουμε μεγάλους όγκους ε, και φυσικά αυξάνεται ο χρόνος των συμβάσεων επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις στις συμβάσεις. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό πώς θέτεται τις επιδόσεις και την απαλλαγή στη συνέχεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν οι απαλλαγές ε, αποτελούνταν και από διαδικασίες αφαιραγκαιότητας σε σχέση με κάποιους δικαιούχους, όμως ε, δεν προσπάθησαν ε, να κάνουν ανάκτηση των πληρωμών που είχαν γίνει στους δικαιούχους αυτούς μέχρι τη στιγμή που χρειαζόταν. Βλέπουμε λοιπόν τέτοια τυπικά προβλήματα και τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε κλασικές περιπτώσεις. Μία ήταν Twitter, όπου αναβλήθηκε η απαλλαγή επειδή υπήρχαν αλλαγές στη διοίκηση και λόγω της ανάγκης να διατηρήσουμε ε, κάποια ορόσημα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, για ε, το σύνολο των οργάνωσης των κοινοπραξιών. Και είχαμε και άλλη μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου αναβλήθηκε η απαλλαγή στην, επί... στην περίπτωση του Artemis Eniac, σημερινό Excel, είχαμε συγχώνευση των δύο κοινοπρασιών ε, στο μέσο ε, του οικονομικού έτους, του λογιστικού έτους. Έτσι λοιπόν είχαμε πολύ λίγο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν ε, συγκεκριμένα στοιχεία για τη διαδικασία της επαλλαγής. Αυτές είναι λοιπόν χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Και για να σας δώσω μια ιδέα για το σύνολο της εύρωστης διαχείρισης, φυσικά ε, έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, τεχνολογική πρόοδος, ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα επιθεωρήσουμε, κυρίως σε ό,τι αφορά την ε, ορθή διαχείριση των επιδόσεων. Δηλαδή, πώς μπορείς να αξιολογήσεις τις επιδόσεις αν εργάζεσαι σε κάτι που θα είναι έτοιμο το 2030. Ο σε καθορισμός των λαθών ή της μη παρουσίασης αποτελεσμάτων ή αποδόσεων ε, δεν ε, προσκαπτεί τη φύση ε, της διαδικασίας. Μερικές φορές τα αποτελέσματα, οι αποδόσεις μπορεί να προβλεφθούν μόνο και με κάποιες πιθανότητες στην καλύτερη περίπτωση, αλλά δεν μιλάμε για σίγουρα αποτελέσματα. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα, οι επιδόσεις των κοινοπραξιών ε, και η εύρωστη διαχείριση εξαρτάται μόνο όχι από τα διάφορους βαθμούς επιτυχίας του προγράμματος έρευνας, αλλά και από τα πορίσματα που μερικές φορές είναι αδύνατον ε, να βρεθούν. Στη σημερινή κατάσταση, αυτό που μπορεί να ειδωθεί κάποια στιγμή ως απώλεια πόρων, μπορεί να θεωρηθεί ως μια επένδυση για μελλοντικά επιτεύγματα. Επομένως είναι πολύ δύσκολη ισορροπία εδώ. Και μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή εδώ που σχετίζεται με τις ε, κοινοπραξίες είναι η απαραίτητη ενεργοποίηση ε, ξένου κεφαλαίου που μπορεί εύκολα να ξεπεράσει ακόμη και την αρχική επένδυση. Ε, των Ευρωπαϊκών Κονδύλιων. Ε, τώρα εδώ μιλάμε για μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις, συνεισφορές που μπορούν να υπάρξουν. Έτσι λοιπόν, οι δραστηριότητε των κυριοπραξιών όχι μόνο ενδυναμώνουν την ευρωπαϊκή μα οικονομία, αλλά φυσικά είδατε, εργαζόμαστε στο θέμα των πυρηνικών, των φαρμάκων, καλύτερα αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν επένδυση για μια καλύτερη ζωή, σε μια καλύτερη ζωή όλων των πολιτών. Αυτό είναι λοιπόν σχεδόν αδύνατο να εκφραστεί με αριθμητικά στοιχεία ή με αξία ή με ποσότητα. Γι' αυτό λοιπόν η διαδικασία της απαλλαγής είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να έχετε πολύ ικανά μέλη της Επιτροπής αλλά για να αναλαμβάνουν αυτά τα καθήκοντα. Είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε νομίζω θίξει όλα τα βασικά θεμελιακά στοιχεία της διαδικασίας της απαλλαγής. Έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, κριτική. Όχι, καλώς. Τότε βλέπω στην ημερήσια διάταξη την συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο, τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, την ε, ε, οργάνωση κατά πολέμηση των απατών. Εμείς έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δαπανώνται και απανταχού του κόσμου να ελέγχονται και από τα εθνικά κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια να δείξουν ενδιαφέρον δηλαδή για το τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτό μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να μας πείτε και εσάς τι σας ενδιαφέρει ε, που θεωρείτε ότι μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Και δεν επιτρέπεται να το θεωρήσετε ως εντό εισαγωγικών προδοσία της πατρίδας εάν εντοπίσετε σφάλματα και τα καταγγείλετε. Και χωρίς τη συνεργασία μαζί σας και εμείς δεν μπορούμε να βελτιωθούμε. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση προς εσάς όλες και όλους να μας βοηθήσετε για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στους ελέγχους. Δεν είναι πάντοτε απλό, διότι βέβαια τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετά μπορεί να συνεπιφέρουν κυρώσεις, ε, μπορεί να σημαίνουν κάποιες απώλειες. Εάν τα βρούμε εμείς, τότε ούτως ή άλλως θα υπάρξουν αυτά, αν βρούμε εμείς τα σφάλματα δηλαδή. Αν τα βρείτε εσείς, τότε μπορούμε να δούμε και τι θα γίνει τα συστήματα διαπίστωση των σφαλμάτων, αν δεν λειτουργούν επιτόπου, τότε το πρόβλημα είναι κοινό και δικό σας και δικό μας. Και το ζήτημα της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για μας είναι κρίσιμη. Στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 28 πάρεδροι, αλλά και 900 πρόσωπα τα οποία εργάζονται για τις υπηρεσίες αυτές. Η συνεργασία όλων αυτών είναι πολύ σημαντική. Τι ελέγχει τώρα το ελεγκτικό συνέδριο, για παράδειγμα, στα διαρθρωτικά ταμεία. Από το 2015 είχαμε 1.081.386 διαρθρωτικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτά ελέγχθηκε 1,1% επιτόπου στις χώρες μέλη. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ελέγξει το 0,02% όλων αυτών των έργων. Το ελεγκτικό συνέδριο επίσης το 0,02%. Και δεν ξέρουμε καν εάν ελεγκτικό συνέδριο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ελέγξει ακριβώς τα ίδια έργα. Γι' αυτό και θέλω να σας ευαισθητοποιήσω η περιοδικότητα, η τακτικότητα των ελέγχων δεν είναι υψηλή. Όμως, σφάλματα μπορεί να διαπιστωθούν καμιά φορά μόνο εάν γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι. Και πρέπει η διαχείριση να γίνεται σωστά, διότι δεν έχουμε περιθώρια, ούτε εσείς ούτε εμείς, να χάσουν την αξιοπιστία τους τα ευρωπαϊκά κονδύλια στα μάτια του κόσμου πρέπει να είναι εγγυημένη η σωστή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γι' αυτό για μας η δράση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και το γεγονός ότι καταφέρει να ελέγξει μονάχα 0,02% όλων των έργων, αντιλαμβάνεστε πού βρίσκεται με τρόπο αυτό το πρόβλημά μας. Πρέπει να γνωρίζουμε αν τα συστήματα αναφορών για να γίνει αυτό πρέπει να μπορούμε να επαφιέμεθα στις χώρες μέλη, στις κυβερνήσεις σας, στα ελεγκτικά σας συνέδρια. Μπορούμε να βασιστούμε στους θεσμούς αυτούς, μπορούμε να βασιστούμε στα εθνικά κοινοβούλια. Εμείς είμαστε οι δύσπιστοι, αλλά νομίζω ότι έχει αποδείξει την αξία της η αυτή. Έχουμε και το γραφείο καταπολέμηση των απατών. Έχουμε πολλά checks and balances μέσα στους μηχανισμούς μας. Αλλά είναι μεγάλα τα ποσά που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως τα κονδύλια αυτά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για πολλούς που έχουν κακούς σκοπούς. Κάθε περίπτωση απάτης την οποία δεν καταφέρνουμε να διαλευκάνουμε, δεν καταφέρνουμε να διαπιστώσουμε, είναι απάτη σε βάρος του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Και όλοι υφιστάμεθα μετά τις επικρίσεις και τη δυσπιστία του κόσμου. Πέρα τώρα της εργασίας αυτής, με την δήλωση αξιοπιστίας, ε, τα ποσοστά σφάλματος, τις απαλλαγές, τις ε, συστάσεις για απαλλαγές που κάνει η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και εν τέλει ολόκληρο το Κοινοβούλιο, χρειάζεται σε κάθε όργανο να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τι γίνεται με τα χρήματα των φορολογουμένων. έχω την εντύπωση ότι από του ελέγχου που έχουμε κάνει ότι οι άνθρωποι κάνουν σωστά τη δουλειά του. Για το ζήτημα τώρα τη καταπολέμηση των απατών, θέλω να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι το γραφείο που έχουμε, όλα αυτά, δηλαδή, με 500 συνεργάτε όλου και όλου, η δουλειά που μπορεί να κάνει δεν είναι παρασταγώνα στον ωκεανό. Χρειάζεται διαρκή βελτίωση των δραστηριοτήτων του γραφείου Αύριο διαθέτουμε ολόκληρη την συνεδρίασή μας στη βελτίωση των διαδικασιών και του τρόπου εργασία του Γραφείου Καταπολέμησης των Απατών. Για μας είναι σημαντικό θέμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να το αφήσουμε να γίνει ένα απλό φιλοσικής. Χρειάζεται να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Το γραφείο Όλαφ λοιπόν είναι για μας σημαντική υπόθεση, διότι είναι και νέο όργανο με την έννοια ότι είναι η ιστορία του μονάχα μιας εικοσαετίας. Ο Όλαφ ε, δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει εξουσία να διεξάγει ποινικέ έρευνες, μόνο διοικητικέ. Δηλαδή μπορεί να ελέγχει λογαριασμούς. Επομένως, για τα περαιτέρω εξαρτάται από τη συνεργασία με τις εθνικές αστυνομίες και εθνικές δικαστικές αρχές. Η συνεργασία αυτή λειτουργεί καλά. Τώρα ιδρύουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί από το 2020. Πρόκειται για Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία, στην οποία μπορούν, είναι εθελοντική συμμετοχή των χωρών μελών, δεν είναι υποχρεωτική. Για την ώρα έχουν ενταχθεί στην εισαγγελία όλες οι χώρες μέλη εκτός από αυτές οι οποίες έχουν opt-out, δηλαδή Ιρλανδία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία, πάντοτε από την αστυνομική συνεργασία. Μέχρι τώρα δεν έχει μπει η Σουηδία και δυστυχώς η Ουγγαρία και η Πολωνία. Και αυτές οι χώρες λαμβάνουν πάρα, πολλά, πάρα πολύ ψηλά ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα πρέπει νομίζω να έχουμε το θάρρος να πούμε εν τέλει ότι όποια χώρα μέλος δεν μπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα λάβει πλέον ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε χώρες οι οποίες αρνούνται να κάνουν τα δέοντα για την διαπίστωση κάθετος εξυχνίαση άπατων σε βάρος των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Είναι τέλος πάντων ένα μέγα εργοτάξιο και μια διαρκής φροντίδα για μας, διότι οι περιπτώσεις απατών που αποκαλύπτει ο Όλαφ με τη βοήθεια των εθνικών αστυνομικών αρχών, μετά αυτά μπαίνουν σε εκθέσεις τις οποίες αποστέλει στις εθνικές δικαστικές αρχές. Πρέπει όμως να είναι εξασφαλισμένο ότι θα επιληφθούν οι εθνικές δικαστικές αρχές, αρχές των υποθέσεων αυτών. Και έχουμε ελλειπή επεξεργασία, όχι από πλευρά δικαστικών αρχών, διότι, όχι διότι δεν θέλουν να συνεργαστούν, αλλά διότι υπάρχουν προθεσμίες. Όταν περάσουν 36 μήνες μέχρι να δηλωθεί η απάτη η υποψία απάτη στον Όλαφ. Μετά χρειάζονται άλλοι 18 μήνες και μετά πολύ συχνά έχουν παρέλθει οι προθεσμίες παραγραφής. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ε, τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τους ευρωπαϊκούς Ελέγχου, δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό. Έχουμε και πολύ καλέ εμπειρίε μέσα από τις χώρες μέλη της Ένωσης, Έχουμε όμως και εμπειρίες διότι τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια έχουν διαφορετικές νομικές βάσεις πάλι με τη σειρά και διαφορετικές αρμοδιότητες μέσα στις χώρες μελή και στα δικαιϊκά του συστήματα και ιδίως όταν πρόκειται για κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Μπαίνει λοιπόν το θέμα ποιες αρμοδιότητες διαθέτει το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο στη χώρα μέλος αν έχει λίγες αρμοδιότητες ασχολείται περισσότερο με τα εθνικά φορολογικά, με τα ε, ε, χρήματα των εθνικών φορολογουμένων περισσότερο και λιγότερο με τα ευρωπαϊκά. Αυτό είναι από τα διδάγματα που έχω λάβει εγώ από την μέχρι τώρα εμπειρία. Αν θέλουμε όμως να βοηθήσουμε και τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν, πρέπει να δώσουμε στα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια μια στέρεα νομική βάση. Αυτή είναι η παράκλησή μου και προ του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι παρόντε εδώ. Πρέπει να φροντίσουμε σε κάθε χώρα η οποία επιθυμεί να ενταχθεί στην Ένωση να λάβουν τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια σημαντικέ αρμοδιότητε. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα που θέλουν και οι ίδιες οι χώρε σε ό,τι αφορά του ελέγχου. Αυτή είναι η μεγάλη μου επιθυμία και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν την έχουμε εκδηλώσει και εντονότερα. Για τα εθνικά κοινοβούλια, τα εθνικά κοινοβούλια είναι δύσκολοι πελάτε. Εσεί δηλαδή για μα είσαστε δύσκολοι πελάτε. να το πω έτσι, διότι τα εθνικά κοινοβούλια όταν προσφέρουμε τέτοιε διοργανώσει, όπω η σημερινή, να καθίσουμε να σκεφτούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα από κοινού, διαπιστώνουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν προσέρχονται καν. λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Όποιος λαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια τα παίρνει, τα διαχειρίζεται και μετά τέλος. Δεν ενδιαφέρεται πλέον. Ο στόχος μας όμως πρέπει να είναι αυτή η διαδικασία και η διαδικασία μάθησης, πώς μπορούμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς, πώς μπορούμε να ε, προτρέψουμε και τις κυβερνήσεις να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Και πρέπει και τα κόμματα που στηρίζουν τις κυβερνήσεις να μην είναι μονάχα δηλαδή υπόθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης η κριτική στάση απέναντι στις κυβερνήσεις σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όταν βρισκόμαστε επί τόπου σε διάφορες χώρες, σε αποστολή, φροντίζουμε πάντοτε να συναντώμεθα με εθνικούς βουλευτές. Δυστυχώς το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα χρονοδιαγράμματα των εθνικών κοινοβουλίων. Πραγματικό δράμα. Όταν πηγαίνουμε εμεί σε αποστολέ, πάμε είτε διότι ε, μα επιτρέπει το κοινοβούλιο εδώ ε, όταν είναι οι διακοπέ των αποκριών, είτε ε, στη διάρκεια των Χριστουγέννων, είτε λίγο πριν από τι θερινέ διακοπέ, όταν και τα εθνικά κοινοβούλια βρίσκονται σε διακοπέ. Σπάνια λοιπόν μπορούμε να βρούμε κάποιον αρμόδιο βουλευτή με τον οποίο να μπορούμε να συνομιλήσουμε. Αυτό που θέλουμε, που είναι ο πραγματικός σε βάθος διάλογος, δεν έχει πετύχει ως τώρα, βέβαια και λόγω έλλειψη ενδιαφέροντος των Εθνικών Κοινοβουλίων και λόγω ε, μη συντονισμού των χρονοδιαγραμμάτων. Εμείς πάντως έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και εσείς έχετε πράγματα όπου χρειάζεστε τη γνώμη μας, θα χαρούμε πάρα πολύ αν μας προσκαλέσετε και θα, προσέλθουμε, και θα φροντίσουμε να προσέλθουμε και έγκαιρα. Αυτά ήθελα να πω για το θέμα αυτό. Τώρα έχετε εσείς το λόγο εφόσον επιθυμείτε. Ωραία. Από την Αλβανία, η κυρία Τσιλαμέτη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα. Είναι θέματα που δεν ενδιαφέρουν μόνο τον, τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, ενδιαφέρουν όλους εμάς, γιατί όσα κονδύλια δίνονται σε εμάς ε, αφορούν την εκτέλεση των όσων κάνουμε. Και άρα θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται με επιμέλεια. Ξέρετε, βλέπω και εγώ σε κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή και έχουμε μια επιτροπή ανεξάρτητη που σε σχέση με τον δημόσιο κορβανά προσπαθεί να καταγράψει, να παρακολουθήσει τις δαπάνες που γίνονται. Το 2015 τροποποιήθηκε ο σχετικός νόμος και αυτή η Επιτροπή τώρα ε, αξιολογεί τις επιδόσεις του προϋπολογισμού μας. Το Υπουργείο Οικονομικών επίσης εμπλέκεται και παρακολουθεί τι γίνεται όσον αφορά την τύχη των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ακριβώς όπως ε, αναφέρατε κυρία Πρόεδρε, αυτά τα κοινοτικά κονδύλια ε, τη παρακολούθησης και από πλευρά τη Όλαφ. Αλλά και από αυτό που σας ανέφερα το Ελληνικό μας όργανο. Ακριβώς όπως γίνεται και με τα δικά μας κονδύλια, του δικού μας προπολογισμού. Και υπάρχει υποχρεωτική λογοδοσία προς την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οπότε αυτός ο υψηλού επίπεδο οικονομικός έλεγχος προβαίνει σε κάποια αξιολόγηση, αλλά προβαίνει και σε συστάσεις προτάσεις, των οποίων την εφαρμογή ελέγχει και παρακολουθεί. Οπότε πολλές από αυτές τις ε, συστάσεις υλοποιούνται, άλλες δεν υλοποιούνται, οπότε για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο έχουμε μια υποεπιτροπή της Επιτροπής μας η οποία έχει αρμοδιότητα ή ακριβώς την παρακολούθηση του αν εφαρμόζονται οι συστάσεις των δημοσιονομικών οργάνων από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της ε, Αλβανίας. Έγινε η τροποποίηση του δικαίου, όπως σας είπα, και έτσι. Ε, διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες αυτού του ελεγκτικού οργάνου να παρακολουθήσει και τους δημόσιους διαγωνισμούς, προμήθειας. Παλιότερα έλεγχονταν μόνο το κατά πόσον ε, ε, υπήρχε ανάθεση κάποιας προμήθειας στον μειοδοτούντα αλλά δεν υπήρχε καταγραφή και αξιολόγηση ε, του αν πιάνω τόπο τα χρήματα του προϋπολογισμού, κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Επομένως τώρα πιάνω τόπο καλύτερα αυτά τα κονδύλια, έχουμε έργα υποδομών, ε, τελικά δηλαδή ωφελούνται έτσι οι φορολογούμενοι της χώρας ε, επίσης. Η Επιτροπή μας εστιάζεται και στο να διοργανώσει δημόσιες ακροάσεις με όλα τα Υπουργεία της χώρας. Κλητεύονται να προσέλθουν στην Επιτροπή και να συζητήσουμε τι έκαναν σε σχέση με τις συστάσεις αυτής της ελεγκτικής υπηρεσίας. και όποτε διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση απάτης οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στην δικαιοσύνη. Τώρα, όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία που είναι στα θέματα που σήμερα συζητούμε εδώ, στο θεματολόγιό μας, πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις γειτονιάζουσες χώρες. Και επίσης έχουμε κάποια προγράμματα και πασχίζουμε να ωφεληθούν όλοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι και έτσι να υπάρχουν ευμενείς οικονομικές συνθήκες για όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος Γκρέσλε. Κύριε Φιλιππόσκη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σας, Πρόεδρε, ότι η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μόνιμο διάλογο μεταξύ των ε, εθνικών κοινοβουλίων και της δικής σας επιτροπής. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η Σερβία έχει θετήσει τη στρατηγική καταπολέμησης ε, της απότης και των παρατυπιών ε, για τα ευρωπαϊκά κονδυλία για την περίοδο 2017-2021. Και αυτό συνοδεύεται και από ένα σχέδιο δράσης που υθετήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017 σε μια κυβερνητική συνεδρίαση. Κατόπιν ε, της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, η Σερβία έχει ένα γραφείο για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων αυτό λοιπόν αφορά όλα τα κονδύλια που λαμβάνει η Σερβία στο πλαίσιο του IPA, του Μέσου Προταξικής Βοήθειας. Αυτό το γραφείο ελέγχου έχει ενισχυμένες αρμοδιότητες. Και έχουν ε, συγκεκριμένους ελεγκτές, επίσης έχουμε δημιουργήσει τις απαραίτητες δομές για τους ελέγχους E-PART ε, και τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Το 2017 το τμήμα καταπολέμησης της απάτης και των ε, παρατυπιών στον τομέα των ευρωπαϊκών κονδυλίων υλοποίησε τέσσερις διοικητικούς ελέγχους Ένας ε, έλεγχος έγινε με την Όλαφ και οι υπόλοιποι τρεις με τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Οικονομικών για την διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στη συνεδρίαση που έγινε το Δεκέμβριο του 2017 στις Βρυξέλλες μεταξύ των εκπροσώπων της Όλαφ με τους Σέρβους εκπροσώπους συμφωνήσαμε ότι προκειμένου να έχουμε μια ακόμη καλύτερη συνεργασία με την Όλαφ θα έπρεπε να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Όλαφ και αυτό το μνημόνιο θα έπρεπε να ορίζει ποιοι είναι οι τομείς συνεργασίας κατά προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κύριος Μέμετη. Ε, okay, thank you. I'm a gentleman, but it doesn't matter. Uh... Δεν είμαι κυρία, κύριος, αλλά δεν πειράζει. Με τιμά πάρα πολύ το ότι με προσκαλέσατε εδώ και ε, να συμβάλλω και εγώ σε όλα όσα έχουμε συζητήσει. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά θα προσπαθήσω όσο μπορώ καλύτερα να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου για το θέμα μας. Δεν νομίζω είμαστε και τόσο αποτελεσματικοί στην αξιοποίηση των κοινοτικών χρημάτων. Και μιλώ για την ε, Μακεδονία, αλλά πιστεύω το ίδιο σημαίνει για τι άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Τέλο πάντων, δεν είμαι εδώ να μιλήσω για τι άλλε χώρε, αλλά για την Μακεδονία. Δεν νομίζω τα πήγαμε τόσο καλά στην αξιοποίηση των χρημάτων που είναι διαθέσιμα σε σχέση με την διασυνορική συνεργασία ε, αλλά και για κονδύλια που αποσκοπούσαν ε, σε άλλα. Ε, πάντως, όταν συζητήσουμε τη διασυνορική συνεργασία, θα δούμε τι στατιστικά υπάρχουν για να δούμε ότι δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα πάντως στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ακούμε συνεχώς είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν διαδραματίζει κάποιον ρόλο. Καθόλου, όχι μικρό, όχι αμυλίδιο, καθόλου. Και δεν αναφέρουμε μόνο στο κοινοτικό χρήμα, αλλά νομίζω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο στα του εθνικού μας προϋπολογισμού. Μια που έχουμε τόσες υπηρεσίες, έχουμε εκεί τους ερετούς που τις τελεχώνουν, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος από αυτών των υπηρεσιών. Απλώς αναφέρονται ε, και κάνουν κάποιον απολογισμό ετήσιο, αλλά ούτε ψηφίζουμε, ούτε έχουμε λόγο στα των υπηρεσιών αυτών. Εμείς ως Κοινοβούλιο τις έχουμε συγκροτήσει όμως αυτές τις ε, υπηρεσίες και έχουμε και την κρατική υπηρεσία οικονομικών ελέγχων, αλλά δεν γίνονται και πολλά πράγματα σε αυτό το μέτωπο. Με μεγάλη μου χαρά ακούω ότι προσπαθείτε να δώστε μια όθηση στα πράγματα και συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει λέγειν, θα πρέπει να έχει κάποιον έλεγχο, όχι μόνο για το κοινοτικό χρήμα, αλλά και για τα χρήματα του δικό μας προϋπολογισμού, ε, επί των οποίων δεν έχουμε έλεγχο. Και νομίζω ότι σε σχέση με την μη αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιδείξουμε πραγματικά προσοχή. Διότι, δεν ξέρω να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι βαθμία σχηματίζεται ένα δίκτυο προσώπων που έχουν πάρα πολύ προχωρημένους τρόπους για να χρησιμοποιούν για τους λάθους σκοπούς τα κοινωτικά χρήματα και έχουν εμπλακεί και πρόσωπα από τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν είναι ευκολότερο να βγάλει κανείς λεφτά στα Δυτικά Βαλκάνια από ό,τι στα κράτη-μέλη. Ίσως αυτό να είναι η απάντηση. Ίσως αυτό να ισχύει. Πάντως πραγματικά πιστεύω ότι και εσείς και εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι συμβαίνει και το ότι υπάρχουν όλα αυτά τα δίκτυα. Ξέρουμε καλά τι γίνεται τι κάνουν. Πάντως δεν έχω τον τρόπο, δεν έχω αρκετά στοιχεία για να τους σταματήσω. Μιλούμε για πρεσβείες που εκπροσωπούν ε, κράτη-μέλη ε, ή μιλούμε για κάποιους εκτός των ε, πρεσβειών. Εγώ σας τα λέω από τα δόντια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σχέση με αυτά. Επομένως θα πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα. Και αυτό το οποίο προτείνεται οπωσδήποτε θα πρέπει να το κάνουν τα εθνικά μήλη. Να αποκτήσουν ουσιαστικό λέγει έλεγχο επί των χρημάτων που σας ανέφερα κοινοτικών και μη. Ευχαριστώ πολύ. Θα λάβουμε υπόψη τα πράγματα αυτά που λέτε όταν θα εξετάσουμε ορισμένες, πολλές από τις χώρες αυτές. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Γαντάγιο από το Κοσυφοπέδιο. Συγγνώμη αν κάνω λάθος τα ονόματά Σα Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη σημερινή συζήτηση. Έχουμε παρακολουθήσει τις ε, εξελίξεις όλα αυτά τα οποία σήμερα αναφέρθηκαν σε σχέση με τις εξελίξεις, με τις διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου. Ξέρετε, στο κρίσιμο πεδίο έχουμε ένα πλεονέκτημα. Έχουμε θεσπίσει νομοθεσία που ευθυγραμμίζεται απολύτως με το κοινωτικό κεκτημένο. Όλοι μας οι νόμοι διέπονται από αυτήν την συμβατότητα. Το ίδιο ισχύει για τον προπολογισμό, το ίδιο ισχύει για τις αρμοδιότητες και λοιπά για τα δημόσια οικονομικά. Η δε εθνοσυνέλευσή μας έχει σχετικές αρμοδιότητες και προβαίνουμε σε ακροάσεις με όλους τους δικαιούχους σε σχέση με τον προϋπολογισμό Είναι τρίμηνη προθεσμία υποβολής ε, έκθεσης σε σχέση με το τρόπο ανάλωσης των κονδυλίων του προπολογισμού. Αυτή η έκθεση επίσης συζητείται στην Εθνοσυνέλευσή μας και κάποια στιγμή εγκρίνεται εάν θεωρείται ότι είναι εντάξει ή απορρίπτεται εάν συμβαίνει το αντίθετο. Από την ίδρυση του κράτους μας συναντήσαμε μια εθνική ελεγκτική υπηρεσία, ε, το Σύνταγμα προβλέπει την ανεξαρτησία της και λειτουργεί αντίστοιχα. Επομένως ανέκαθεν να από ανεξαρτησία στη λειτουργία της αυτή η υπηρεσία και σε τακτά διαστήματα ασκεί οικονομικό έλεγχο σε όλα τα δεσμικά όργανα του κράτους μας που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό. Ε, αυτό το δεσμικό όργανο ασκεί τον οικονομικό έλεγχο επί όλων των κρατικών υπηρεσιών όπως είπαμε που σχετίζεται με τον δημόσιο κορβάνα. Είναι αυτό μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη νομίζω ότι είναι θετικό το ότι το 2009 συγκροτήσαμε μια επιτροπή. Αυτή η δική επιτροπή έχει μόνη αρμοδιότητα την παρακολούθηση των δημοσίων οικονομικών. Και αυτή η επιτροπή ελέγχει τις εκθέσεις των ελεγκτών και τις εκθέσεις σε σχέση με τις επιδόσεις της, σε επίπεδο οικονομικό. Τα συμπερασματά της συζητούνται στο Κοινοβούλιο, είναι αντικείμενο έγκρισης με ψηφοφορία. Μόνος έχει σημαντικό ρόλο στην δημοκρατία μας αυτή η Επιτροπή. Και παρακολουθεί τι τα κονδύλια του προϋπολογισμού. αυτά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Θεωρώ ότι είναι καλής ποιότητας ο έλεγχος που ασκούμε στα δημόσια οικονομικά. Παρ' όλα αυτά,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 Ε, μελετήσαμε την έκθεση σε σχέση με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες ε, και επίσης σε σχέση με την λειτουργία των υπηρεσιών που λειτουργούν στα κράτη, κράτη-μέλη. Πάντως, Όσον αφορά την Ιούλεξ, την ε, αποστολή ε, της ε, Ένωσης που είχε αναλάβει τη συγκρότηση του κράτους μας, για το κράτος δικαίου κλπ. Έκθεση για τη Ιούλεξ δεν έχει γίνει. Βεβαίω και θα έπρεπε να έχει θωρακιστεί από πολιτικές επιρροές και παρεμβάσεις το κράτος δικαίου στη χώρα μας η δικαστική εξουσία βέβαια ετύχανε κάποιου είδου προστασία από την αποστολή Γιούλεξ Οπότε γι' αυτό υπάρχουν κάποια, κάποια όρια στο πόσο ωφελήθηκε η χώρα από τα κοινωτικά κονδύλια και από την αποστολή Γιούλεξ. Οπότε γι' αυτό και σας ερωτώ, έχει ποτέ προβεί σε κάποιο είδους απολογισμό Γιούλεξ για το πώς ανέλωσε τα κοινωτικά χρήματα στο Κόσοβο. Και έχω μελετήσει την έκθεση που σας είπα του κυρίου Πέτρη που αφορούσε ε, την κατάσταση αυτή και θέλω ε, ο κύριος Σασαρβαμάς την έκθεσή του, για την έκθεσή του να μας ε, μιλήσει περισσότερο. Και όντως θα πρέπει να δούμε εάν το χρήμα πήγε εκεί που έπρεπε. Εκεί που όφιλε να πάει. Σας ανέφερα την δικαιοσύνη, αλλά αφορά αυτό και άλλες πτυχές της λειτουργίας του κράτους μας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Ευχαριστώ και για την ερώτησή σας. Έχουμε δουλέψει πολύ για τα θέματα της EULEX και η Επιτροπή μας πήγε τουλάχιστον δύο φορές στο Κόσοβο τα τελευταία 15 χρόνια, συνολικά τρεις φορές. Και εγώ μάλιστα συμμετείχα μια φορά σε σχετική αποστολή και έχουμε ασχοληθεί όπως είπα σε βάθος με την EULEX. Αυτό που λέτε δεν με χαροποιεί σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της EULEX Ασχοληθήκαμε βέβαια και με τις καταγγελίες σε βάρος της Ulex. Τη συζητήσαμε και με τη δική μας εδώ Επιτροπή Εξωτερικών. Ε, υπήρξε και σχετική έκθεση. Οι εκθέσεις που υποβάλλει η Ulex απευθύνονται στην Επιτροπή Εξωτερικών. Όμως, μετά από τα όσα μας είπατε, θα το κάνουμε θέμα εμείς εδώ. Και σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις μας μετά τις θερινές διακοπές θα ζητήσουμε να ενημερωθούμε και αν αυτά που λέτε είναι πράγματι σωστά. Είναι μια αποστολή μεγάλη, αποστολή δαπανηρή, μιλώ για την EULEX, με πολύ προσωπικό και θα είναι πολύ δυσάρεστο εάν η αντίληψη που έχει ο κόσμος εκεί είναι ότι προκαλεί δυσκολίες. Γι' αυτό λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την υποδείξή σας και θα σας ενημερώσουμε και για το τι, έχει, θα έχει προκύψει δηλαδή από τις αυτές. Αν έχετε στατιστικές, εκθέσεις, προφορίες, σας παρακαλώ να μας, τις, να μας τις διαβιβάσετε. Ή δυνατόν βέβαια στα αγγλικά. γιατί έχουμε μια δυσχέρεια να μεταφράζουμε γλώσσες εκτός των γλωσσών των χώρων μελών. Πολύ ευχαριστώ πάντως θα εγκύψουμε στο θέμα αυτό που θέσατε υπόψη μας. Έχει περάσει μια διετία που δεν ασχοληθήκαμε πλέον με την EULEX, αλλά έχουμε αφορμή από αυτά που λέτε να επανακαμψούμε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Ας περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ακρόαση αν δεν έχετε άλλο τίποτε να πείτε. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κυρίους Τσέλερ και Κλίντς για να κάνουν τις σχετικές εισαγωγικές τοποθετήσεις τους. Ο κύριος Κλίντς πρώτα. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευρωβουλευτή Κλίν από την ομάδα των Φιλελευθέρων. Προτιμάς να αρχίσεις εσύ κύριε Σάβαμα. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί την προϋπόθεση για καλές γειτονικέ σχέσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι πολιτικές καταστάσεις η πολιτική κατάσταση μάλλον της περιοχής γίνεται σιγά σιγά πιο σταθερή και ότι έτσι ανοίγονται και οικονομικές δυνατότητες και ευκαιρίες. Για να τα πετύχουμε τα πράγματα αυτά χρειάζεται βέβαια μια σχέση εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται με νομοθετικά μέτρα, αλλά διαμορφώνεται μέσα στην πάροδο του χρόνου και όταν βλέπει ο κόσμος ότι η συνεργασία αποδίδει καρπούς για όλους, όχι για τη μια πλευρά μόνο, αλλά για όλους τους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες. Αυτό ισχύει ιδίω για την περιφέρεια των Δυτικών Βαλκανίων, ακόμη περισσότερο. Και γι' αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω τις και τους εκπροσώπους των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για τις τοποθετήσεις τους. Εγώ προσωπικά γνωρίζω μόνο την Αλβανία, καμία από τις άλλες ενδιαφερόμενες χώρες και γι' αυτό είναι σημαντικό και ενδιαφέρον για μένα που ακούω προσωπικές αναφορές από τους συμμετέχοντες και μου δίνουν μια εικόνα για την κατάσταση των χωρών τους. Χώρες οι οποίες για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεγάλη σημασία, διότι συναποτελούν μέρος της Ευρώπης. Αν δούμε το κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και ο τελευταίος του όροφος δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένος, δείχνει καθαρά ότι, με τον τρόπο αυτό συμβολικά ας πούμε, ότι και η Ευρώπη δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό μου θυμίζει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που ακόμα δεν έχουν γίνει μέλη της Ένωσης. Όμως, μέσο και μακροπρόθεσμα έχουν το στόχο να ενταχθούν. Όμως αυτό το στόχο θα τον επιτύχουμε μόνο αν οι χώρες αυτές μπορέσουν να προσεγγίσουν βήμα-βήμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν βήμα-βήμα υιοθετήσουν τις αξίες πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι μονάχα ελευθερία, ειρήνη και ευημερία, αλλά και το δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοεί αυτήν ως χώρο δικαίου και γι' αυτό πρέπει να υλοποιηθεί και αυτή η διάσταση και για τις χώρες αυτές. Οι έξι εμβληματικές πρωτοβουλίες, flagship initiatives της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν και στόχο τη δημιουργία κράτους δικαίου. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία που λέγεται ε, Πρωτοβουλία Ενίσχυση του Κράτους Δικαίου. Η σημασία αυτής τη πρωτοβουλίας είναι πραγματικά τεράστια. Εμείς ζητήσαμε μελέτη για την ορατότητα των διαμεθοριακών και διεθνικών συνεργασιών. CBC, Cross Border Cooperation δηλαδή στα αγγλικά, μέσα στα πλαίσια του μέσου για την προενταξιακή στήριξη. Και ευχαριστώ εδώ του συντάκτες της μελέτης, Άκερμαν και συνεργάτες, και τους άλλους ε, βεβαίω συναρμόδιους, όπως και τον Ευρωβουλευτή κύριο Τσέλερ. Από, τις, από το περιεχόμενο της μελέτης φαίνεται που βρισκόμαστε. Δεν είναι πάντοτε απλό, να δει κανείς και να μπορέσει να αξιολογήσει το μέτρο στο οποίο έχουν επιτευχθεί έω τώρα οι στόχοι. Παρ' όλα αυτά, δείχνει η μελέτη και τι έχουμε επιτύχει και πού βρισκόμαστε τώρα και δείχνει επίσης ότι και τα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί για τους σκοπούς αυτούς, δηλαδή αυτά τα προενταξιακά κονδύλια, ότι αυξάνονται διαρκώ από, τη μία μεσοπρόθεσμη, από τον ένα μεσοπρόθεσμο μάλλον σχεδιασμό στον άλλο. Και για το 2020 2027, που δεν έχει εγκριθεί τελειωτικά ακόμα, προβλέπεται ένα ποσό της τάξης των 14 και μισό δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για πρόοδο λοιπόν και με την έννοια αυτή είμαι και εγώ αισιόδοξο ότι θα επιτύχουμε συστηματικά να φέρουμε τις χώρες αυτές όλο και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο είναι σημαντικό διότι στο μεταξύ η περιοχή αυτή έχει γίνει στόχος φιλοδοξιών και άλλων φορέων και άλλων χωρών. Τουρκία, χώρες του Περσικού κόλπου, Ρωσία, ακόμα και οι Κινέζοι φαίνεται, σύμφωνα με πολλούς, ότι έχουν ανακαλύψει το δυναμικό της περιοχής αυτής. Έχουμε λοιπόν ενδιαφέρον ιδιαίτερο εμείς η Ευρώπη των 28, όπως στο μέλλον θα είμαστε η Ευρώπη των 27, να φέρουμε τις χώρες αυτές όσο γίνεται πιο γρήγορα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έκανα βέβαια ένα μικρό σφάλμα προηγουμένω, γιατί συνεισηγητή σα είναι ο κύριο Τσέλερ. Αυτό θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Τσέλερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο συνάδελφό μου Κλίντ μόλι πριν. εάν θέλουμε, όταν βρισκόμαστε μάλλον στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, βλέπουμε μεγάλη προθυμία των πολιτών να ενταχθούν οι χώρες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν φτάσει ορισμένοι να μιλούν και για ανυπομονησία σε ό,τι αφορά την πορεία της, των χώρων αυτών προς την ένταξη. Βέβαια, οι συνθήκες είναι αυτές που είναι. Και η πρόεδρος μας ήδη στην αρχική της τοποθέτηση εξήγησε ότι για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν κριτήρια, τα λεγόμενα κριτήρια της Κοπενχάγης, τα οποία με την ευκαιρία επιθυμώ να υπενθυμίσω. Από το 1995 ισχύουν τα κριτήρια αυτά, τα οποία εγκρίθηκαν και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται πρώτο-πρώτο και θεμελιώδες το κριτήριο της θεσμικής σταθερότητας ως εγγύηση για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, προστασία των μειονοτήτων. Δεύτερο κριτήριο. Δημιουργία λειτουργικής οικονομίας της αγοράς. Τρίτο κριτήριο, η ικανότητα πλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους και για την υιοθέτηση του λιγόμενου κοινοτικού και κτημένου, δηλαδή όλων των κανόνων και στρατηγικών αποδοχή των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και ιδίως για το τρίτο αυτό κριτήριο κανόνες, πρότυπα, μάλλον περισσότερα γίνονται παρά λιγότερα και αποτελούν σημαντική πρόκληση και για τις χώρες μέλη της ίδιας ό,τι αφορά την εφαρμογή τους. Για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων πρέπει ωστόσο μια χώρα τουλάχιστον να ανταποκρίνεται στο πρώτο κριτήριο, δηλαδή κράτος δικαίου, δημοκρατία, σεβασμό ανθρώπινων δικαιωμάτων, προστασία μειονοτήτων. Τώρα, για το πόσο έχει προχωρήσει η διαδικασία που κατευθύνει προς την ένταξη, αυτό μας το δείχνουν οι αιτήσει εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα κέριο σημείο εδώ είναι πάντα η αποτίμηση για το κατά πόσο η κατάχρηση κρατικών κονδυλίων, η, η διαφθορά αν θέλετε διαφορετικά, έχει ανακοπεί ή εν πάση περιπτώσει αν έχει καταπολεμηθεί δραστικά, ώστε τα δημόσια κονδύλια είτε του ντόπιου φορολογούμενου είτε του ευρωπαίου φορολογούμενου εφόσον πρόκειται για ενισχύσεις που προέρχονται από την πολιτική γειτονία ή από την προενταξιακή στρατηγική, αν προστατεύονται. Εάν δαπανώνται σύμφωνα με τους συγκεκριμένου σκοπούς τους και όχι για να πάνε στις τσέπες των διαφόρων. Και εδώ οφείλω να πω ότι ναι, μεν έχουν γίνει κάποια, κάποια βήματα πρόοδου στι διάφορε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικέ προκλήσει, δηλαδή κυρίω την καταπολέμηση τη διαφθορά. Είχα πει προηγουμένω ότι το θέμα αυτό σημαίνει και ειδική στόχευση στην διαμεθοριακή συνεργασία. Ιδίω διαμεθοριακή συνεργασία μεταξύ περιφερειών και όπως είπα, ανέφερα και την ανυπομονησία πολλών πολιτών, ιδίω τη νέα γενιά, την οποία κατανοούμε, αλλά από την άλλη μεριά οφείλουμε να επιμείνουμε στον σεβασμό και πλήρωση των κριτηρίων. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βελτίωση της συνεργασίας, όπως είπα και αρχικά, εδώ δραστηριοποιούνται τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για μια βελτιωμένη διαμεθορική συνεργασία στα πλαίσια της ε, Περιφερειακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Έχουν διευρυνθεί τα σχετικά νομικά εργαλεία, έχουν εξασφαλιστεί με νέους κανονισμούς και εγώ θα ταχθώ υπέρ της ιδέας να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή και όχι μονάχα πάντοτε να αναμένουμε την πολιτική διαδικασία της ένταξης που βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστεί αλλά ας μην είμαστε όλοι υπεραισιόδοξοι. Ακούμε τώρα για το έτος 2025, όπου ενδεχομένως κάποιες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να ενταχθούν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η ένταξη θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στην προένταξη διαδικασία. Αν θα είναι τώρα το 2025, ίσως νωρίτερα ή ίσως αργότερα, αυτό θα φανεί σιγά και με τον καιρό. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν για ενισχυμένη συνεργασία. Ο συνάδελφός μου Κλίντς θύμισε ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι προσπαθούν να προσελγίσουν στις σφαίρες επιρροής τους στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσα στα πλαίσια μιας νέας παγκοσμιοποιημένης πολιτικής. Το θέμα βεβαίως είναι και δικό σας, αξιότιμες κυρίες και κύριοι των, ε, κοινοβουλίων, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ποιο δρόμο θέλετε να ακολουθήσετε τον πιο κοπιαστικό δρόμο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να ακούσετε το άσμα των σιρήνων άλλων που ίσως σας προσφέρουν κάποια οικονομικά πλονεκτήματα. Κύριε Άκερμαν, έχετε το λόγο για την παρουσίαση της μελέτης. Thank you. Um... Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να βλέπετε την παρουσίασή μου. Mm. Ωραία, πρόκειται για μία ενημέρωση. Όχι μελέτη, είναι κάτι διαφορετικό. So, um, yes, the objectives of the, uh, Οι στόχοι της ενημέρωσης για να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα και την προβολή τη ε, χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια επικεντρώνονται συνήθω στη και συνεργασία. Θα πρέπει να τονίσω ότι δεν πρόκειται για μια αξιολόγηση, ούτε μια κριτική των επιδόσεων. Η έρευνα εξακολουθεί να συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε νέα έγγραφα που λαμβάνουμε από την ΚΑΠΑΔΕΛΤΑ ΝΙΑΡ και από άλλες πηγές. Και όπως ανέφερα στην αρχή, καθώς πρόκειται για μια ενημέρωση παρά για μια μελέτη, έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογή και περιορισμένο προϋπολογισμό. Και επομένως η έρευνα έγκυται σε συνεντεύξεις ε, που ελήφθησαν από ένα μικρό αριθμό στρατηγικών ενδιαφερομένων μερών από τη Γενική Διευθυνσία, τις αντιπροσωπείες στα Δυτικά Βαλκάνια και κάποιες διαχειριστικές αρχές από τα κράτη-μέλη όπου υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία, προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και το Interreg. Δημοσίες ε, Δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες αξιολογούμε, όπως κατευθυντήρες γραμμές, εκθέσεις αξιολόγησης, ε, θέματα που αφορούν ε, την προβολή κτλ. Θα σας παρουσιάσω μια επισκόπηση της χρηματοδότησης συνολικά για το πρώτο γύρο του Μέσου Πρόταξης Βοήθειας 2007-2013 ε, είχαμε ένα συνολικό ε, ποσό 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, για το δεύτερο ε, IPA. Η εκταμίευση ήταν 11,7 ε, δισεκατομμύρια. Τα εθνικά προγράμματα καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία αυτή της της εκταμίευσης ε, περίπου το 75%. Το 70%. Σε ό,τι αφορά τώρα στα Δυτικά Βαλκάνια, τα εθνικά προγράμματα ε, φτάνουν στο 4, στα 4 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης. Τα περιφερειακά προγράμματα συμπεριλαμβανομένες και της ε, Τουρκίας καλύπτουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ και Συγκεκριμένα, η διασυνορική συνεργασία μεταξύ των χωρών IPA στα Δυτικά Βαλκάνια φτάνει στο ποσό των 83 εκατομμυρίων. Για το EPA1, για σκοπούς σύγκρισης, φαίνεται σαν ε, η διασυνοριακή συνεργασία ε, να μειώθηκε ως προς τους πόρους, ε, γιατί είχαμε 33 εκατομμύρια ε, που δόθηκαν σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που αφορούσαν και την Κροατία, ενώ το συνολικό ποσό ήταν 93 ε, εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν, αν συγκρίνουμε με το ΙΠΑ 2, ε, που έχουμε 83 εκατομμύρια, στο ΙΠΑ 1 μας μένουν 64 εκατομμύρια για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Δύο κύρια θέματα της διασυνοριακής συνεργασίας ε, που καλύπτονται είναι ο τουρισμός, ε, η πολιτιστική κληρονομιά, περιβαλλοντική προστασία, ανεργία και ε, κοινωνική ένταξη. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι είχαμε σημαντικές εξελίξεις από το ΙΠΑ 1 στο ΙΠΑ 2. Συγκεκριμένα Τώρα υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει διάφορες κατευθυντήρες γραμμές και συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Υπάρχει επίσης και καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ του μέσου περιοδοξικής βοηθείας και των εθνικών πολιτικών στο στάδιο προγραμματισμού η θεματική εστίαση κάπως έχει μετριαστεί. Ε, αυτό θέλει να διευκολύνει την κατανόηση για το πώς η στήριξη αυτή μας οδηγεί σε αλλαγές. Ό,τι αφορά τώρα την προβολή, σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι σαφές από διάφορα έγγραφα και κατευθυντήριες γραμμές και από συζητήσει με τα διαφερόμενα μέρη ε, από ανθρώπου με του οποίου συζητήσαμε, από τη ΓΑΜΑ Δελτανίρ και από τις αντιπροσωπείες στα Δυτικά Βαλκάνια. Επομένω, οι κύριες αλλαγέ ε, που έκαναν μια μεγάλη διαφορά για τη διασυνορική συνεργασία σχετίζονται με την απλούστευση της διαχείρισης. Συγκεκριμένα, μια διαχειριστική αρχή υπάρχει τώρα για κάθε πρόγραμμα διασυνορικής συνεργασίας και οι εταίροι στις ε, όμορες χώρες υποβάλλουν μία και μόνη αίτηση και εκθέσεις πρόοδου. Δεν ε, υπάρχει λοιπόν ε, επικάλυψη με το τι κάνουν οι αρχές στις χώρες εταίρους. Είναι πολύ δύσκολο στα πλαίσια μιας τόσο σύντομης παρουσίασης να σας παρουσιάσω όλες τις εξελίξεις. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε εδώ αυτά που θεώρησαν κατά την άποψή μας τα διαφοράμενα μέρη ως κύριες εξελίξεις. Ίσως είναι σημαντικό να σκεφτούμε για μια στιγμή τι εννοούμε όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα. Είναι ο βαθμός στον οποίο τα προγράμματα παράγουν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ορίζονται στον κανονισμό 236 του 2014 ως ε, η, τα output, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος. Τα αποτελέσματα δεν ορίζεται μάλλον αυτό, όπως γνωρίζω. Ε, είναι λοιπόν τα αποτελέσματα βιώσιμες αλλαγές στις επιδόσεις, στις τάσεις, στη συμπεριφορά και στις αντιλήψεις κάποιων ομάδων στόχων και στους θεσμούς, τα συστήματα κτλ. που λαμβάνουν ε, οικονομική στήριξη από την Ένωση τα output δεν αντικαθιστούν τα αποτελέσματα. Είναι απαραίτητα για την επίτευξη των αποτελεσμάτων, αλλά χωρίς ε, τα αποτελέσματα δεν ε, μπορούμε να σας πούμε τι έχει αλλάξει στην πραγματικότητα ως αποτελέσμα της παρέμβασης. Και υπάρχει περιορισμένη έρευνα για τον αντίκτυπο, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να το συλλάβουμε. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στα αποτελέσματα και στις βιώσιμες ε, αλλαγές σε ό,τι αφορά την αλλαγή των συμπεριφορών και των στάσεων. Είναι σημαντικό αυτό γιατί σε διάφορα έγγραφα αναφέρονται διάφορα πράγματα. Παραδείγματο χάρη γίνεται λόγο για αποτελέσματα, για αντίκτυπο, για output αποδόσει. Επομένω, είναι ε, σημαντικό να έχουμε ένα συστηματικό ορισμό όλων αυτών των σημείων. Πάντω, τα αποτελέσματα, outcomes, είναι αυτά που μετράνε πιστεύω. Τώρα, Προχωράμε στην προσθεμένη αξία της διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από την Ένωση. Είναι κάτι που ε, θα πρέπει να εξετάσουμε, δηλαδή την αποτελεσματικότητα του μέσου πρωτοεξιακής βοήθειας γενικότερα στο πλαίσιο αυτής ε, της ενημέρωσης. Μας ζήτησαν να επικεντρωθούμε στη διασυνοριακή συνεργασία έτσι λοιπόν για την αποτελεσματικότητα εξετάσαμε την πρόσθετη αξία και τα αποτελέσματα στο οποίο θα φτάσω ένα λεπτό. Δυσυνορία και συνεργασία λοιπόν που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ε, μια σειρά προστιθέμενων αξιών. Έχουμε χρηματοδότηση για περιφερειακές ε, ε, περιοχές που έχουν λίγη πρόσβαση σε άλλα κονδύλια, καλύπτει τα κενά ε, και σε τομείς που έχουν παραμεληθεί, δεν επικαλύπτεται με άλλη χρηματοδότηση, γιατί τα περισσότερα εθνικά προγράμματα τείνουν να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εθνικών θεσμών και συστημάτων επικεντρώνεται σε εύκολους στόχους, δηλαδή ε, καλές ε, σχέσεις γειτονίας, που είναι δύσκολο να μετρηθεί και είναι προσβάσιμο σε εταίρους με μικρότερες ικανότητες, όπως παραδείγματο χάρη, τοπική αυτοδιοίκηση σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μας είπαν ότι το ΙΠΑ 1 βοήθησε να αναπτυχθούν οι ικανότητες των ομάδων αυτών για τη διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Επίσης, ε, είναι ευέλικτο και πραγματικά γίνεται συντονισμός των προϊόντων για να ανταποκρίνονται στις ε, τοπικές ανάγκες. Υπάρχει ηγεσία από την κοινότητα, κάτι που προωθεί την ιδιοκτησία των προγραμμάτων και ε, παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχει μια έλλειψη σύνδεσης με τις εθνικές πολιτικές ε, πέρα από το στάδιο του προγράμματος και αυτό κατά κάποιο τρόπο περιορίζει την προσθέμενη αξία της διασυνοριακής συνεργασίας. Όμως συνολικά το feedback που είχαμε είναι ότι η προσθέμενη αξία είναι ιδιαίτερα εντονή και ισχυρή και συμπληρώνει πολύ καλά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τώρα, για να φτάσουμε στα αποτελέσματα της διασυνοριακής συνεργασίας, δηλαδή τι ακριβώς έχει αλλάξει ως ε, αποτέλεσμα αυτής της χρηματοδότησης στον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι ομάδες μεταξύ τους και που λειτουργούν. Ένα πολύ σημαντικό σημείο ήταν το θέμα της συμφιλίωσης και της ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνης ε, για να ξεπεραστούν ε, ιστορικές εντάσεις ή διαιρέσεις. Έχει, έχει ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των δημοσίων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στο πρώτος γύρος του IPA 2007-2013 ε, ουσιαστικά συνέβαλε στο να βρεθούν μαζί ε, εκδιφερόμενα μέρη που συνήθως δεν θα συνεργάζονταν, ε, προώθησε μια κοινή κατανόηση και δέσμευση στις διασυνορικές περιοχές για θέματα όπως το περιβάλλον, κοινωνικά ζητήματα, πολιτιστική κληρονομιά κτλ. Παρ' όλα αυτά, η αξιολόγηση της διασυνεργικής συνεργασίας που κάλυπτε το EPA 1 προέκυψε με σαφήνεια ότι υπήρχαν πολύ λίγες ουσιαστικές πληροφορίες ως προς τα αποτελέσματα. Αυτή ήταν και η δική μας εμπειρία. Υπήρχαν ε, πολλά παραδείγματα για πράγματα που έχουν αλλάξει, όμως δεν υπήρχε μια συστηματική καταγραφή και ανάλυση και ουσιαστικά έχουμε την αίσθηση ότι αυτά είναι κάποια καλά παραδείγματα που τείνουν να διευρύνονται και να προβάλλονται. Όμως αυτό δεν μας δίνει απαραίτητα μια πλήρη εικόνα. Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε υπερβολή προς τα αποτελέσματα. Όμως δεν υπάρχει μια πλήρης εικόνα στην πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το EPA2, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο εφαρμογή και δεν είναι δυνατόν να πούμε πολλά για τα αποτελέσματα, για το τι πράγματι αλλάζει. Όμω, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ε, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και την αξιολόγησή του. Όμω, ε, στην πράξη, η υποβολή εκθέσεων και ανάλυση θα είναι καλύτερη ή θα υπάρχουν τέτοια παράπονα με την ε, αξιολόγηση του IPA1 και του σκέλους της διασυνορική συνεργασίας, όπου δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες σε σχέση με τα αποτελέσματα για το τι έχει αλλάξει. Τώρα, περνάμε στο θέμα της προβολής. Εξετάσαμε διάφορα έγγραφα και συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2015 που τονίζουν την ανάγκη να βελτιωθεί η επικοινωνία, η κατανόηση και η ευαισθησία, η ευαισθητοποίηση απέναντι στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στις χώρες ε, της διεύρυνσης. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα δεκασέλιδο που παρέχει πληροφορίες για το EPA και καλύπτει τα έτη 2015-16 που θα τρέχει μέχρι το 2020. Αυτό επικεντρώνεται, αναφέρει το θέμα της ε, ευαισθητοποίησης, αλλά επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις δραστηριότητες και στις ε, δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής. Αναφέρει διάφορες δημοσκοπήσεις και έρευνες, όχι όμως ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι η Κομισιόν έχει μία απόρριτη στρατηγική επικοινωνία. δεν μπορούμε φυσικά να την σχολιάσουμε. Και για λόγους που κάπως ε, αναφέρθηκαν προηγουμένως, η γάμα δελτανία δεν έφερε ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Task Force, Task Force όπου μάλλον η οποία συντονίζεται και συνεργάζεται με τη ΓΑΜΑ Και ένα άλλο έγγραφο που έχουμε είναι οι απαιτήσει επικοινωνία και προβολή ε, για του ε, εταίρου που εφαρμόζουν το πρόγραμμα. Επομένως, κατευθυντήριες γραμμές ε, ουσιαστικά μας πρότεινε ένα τρόπο να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων προβολής και επικοινωνίας ε, παρέχοντας αποδείξεις για τις ε, δραστηριότητες προβολής. Όμως αυτό στην πραγματικότητα δεν σου λέει αυτό πόσο αποτελεσματικές ήταν οι δράσεις αυτές, απλώς ότι έγιναν. Λοιπόν, να δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα τι συμβαίνει με την προβολή και τι σημαίνει όταν μιλάμε για προβολή της χρηματοδότησης της συνολικής συνεργασίας της Ένωσης. Υπάρχουν βεβαίως πολλές δραστηριότητες προβολής, ε, τονίζονται ιδιαίτερα όπως σας ανέφερα. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες γραμμές. Θεωρείται ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση σχέση με το EPA1 και σίγουρα είχαμε κάποιες καινοτόμες ε, προσεγγίσεις στρογγυλές τράπεζες ε, όπου συμμετείχαν και οι δικαιούχοι από απομακρυσμένες ε, ε, συνοριακές περιοχές που κάθισαν όλοι από κοινού για να συζητήσουν τις εμπειρίες τους με ε, ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση μάθησης, αλλά και ένας πολύ καλός τρόπος να ενισχύσει την προβολή. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα μας είπαν ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι καλή η προβολή εν μέρη βάσει κάποιων δικτών όπως περνούν το σχάρι ο αριθμός ε, των αιτήσεων για επιχορηγήσεις. Αυτό επιβεβαιώνει την προβολή μεταξύ όσων κάνουν αίτηση, αλλά αυτό φυσικά δεν σου λέει τι γίνεται με την προβολή στο ευρύτερο κοινό, ούτε με το ποιε είναι οι αντιλήψει του κοινού και ποια είναι η κατανόηση της ε, χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται να υπάρχει πολύ λίγη συστηματική έρευνα στο θέμα της δημόσιας ευαισθητοποίησης, της ευαισθητοποίησης του κοινού και της κατανόησης της χρηματοδότησης της διασυνορικής συνεργασίας. Ρωτήσαμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αν μπορούν να μας δώσουν παραδείγματα από δημοσκοπήσεις ή έρευνα στην κοινή γνώμη. Μας είπαν αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες, αλλά νομίζω ότι μόνο σε ε, στις χώρες όπου μιλήσαμε στις αντιπροσωπείε μπορούσε κάποιος να μας δώσει συγκεκριμένο παράδειγμα κάποιας δημοσκόπησης που να επικεντρώνεται συγκεκριμένα στην ε, χρηματοδότηση της συνοριακής συνεργασία. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει κάποια τέτοια δραστηριότητα, απλώς ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε δεν το γνώριζαν αν έχει γίνει ή όχι. Και νομίζω ότι αν δεν γίνονται τις δραστηριότητες είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πόσο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία και η προβολή όσο προς την ευαισθητοποίηση και να μάθουμε αν οι άνθρωποι έχουν ε, ουσιαστικά λανθασμένη κατανόηση. Επίσης αναρωτιόμαστε για αν οι δραστηριότητες για τις οποίες μας μίλησαν επικεντρώνονται κυρίως στις ίδιες συνορικές περιοχές ως προς το αποτέλεσμά τους. Είναι σημαντικό να προτείνουμε να το γνωρίζει αυτό και ευρύτερο πληθυσμό. Δεν είναι σαφές από τις ε, πληροφορίες και τις συζητήσει που είχαμε ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο ότι συμβαίνει. Όπως είπα και πριν, η αξιολόγηση της διασυνορικής συνεργασίας του ΙΠΑ 1 μας έδειξε ότι υπήρχε μια έλλειψη αποτελεσμάτων. Πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Γιατί αν μπορείς να τονίσεις με συγκεκριμένο τρόπο τι έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης, αυτό είναι κάτι πολύ καλό που μπορείς να πουλήσεις παρά να βασίζεσαι σε κάποιες ε, ιστορίες, σε κάποια ανέκδοτα που διηγούνται άνθρωποι που είναι μέρος του συστήματος. Αν ε, μπορείς να αναφέρεις αποτελέσματα που προέρχονται από συστηματική έρευνα, ίσως αυτό να είναι κάτι πιο ισχυρό από το να επαναλαμβάνεις ε, αποδείξεις που προέρχονται από διάφορες ιστορίες. Συμπερασματικά, προτείνουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη να βελτιωθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου. Ο αντικτύπος ε, είναι ε, κάτι πολύπλοκο. Όλοι ε, τα όργανα, όλοι οι θεσμοί ασχολούνται με το θέμα αυτό. Σίγουρα υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι η Κομισιόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς συζητούνται όλο και περισσότερα τα αποτελέσματα. Και ξέρω ότι η Κομισιόν ε, θέλει ουσιαστικά να κατανοήσει περισσότερο ε, το πώς γίνεται η αξιολόγηση και θέλει ουσιαστικά να προωθήσει και την αξιολόγηση και την εκμάθηση στην πλαίσιο της ΓΔΝΙΕΡ. Όμως, χρειάζεται πιο συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, δηλαδή το τι αλλάζει στην πραγματικότητα, το πώς συσχετίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, για το πώς αντιλαμβάνονται ο ένας τον άλλον, για το πώς ε, ε, εργάζονται και συνεργάζονται οι θεσμοί και τα συστήματα. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τη διασυνοριακή συνεργασία, αλλά γενικότερα για τη χρηματοδότηση του μέσου προταξιακής βοήθειας ίσως θα έπρεπε να βασιζόμαστε mm. λιγότερο σε κάποιες αποδείξεις ε, ε, που απλώς κυκλοφορούν ως φήμες ε, και δεν αντικατοπτρίζουν τα βιώματα του πληθυσμού. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε κριτική κοινωνική εκμάθηση. Νομίζω ότι στο παρελθόν η αξιολόγηση έτεινε να βασίζεται στη λογοδοσία, και νομίζω ότι ίσως τώρα πρέπει να... Ε, και μάλλον ε, φαινόταν ότι έκαναν κάποια αξιολόγηση χωρίς να διασφαλίζουν όμως ότι υπήρχε μια διαδικασία εκμάθησης. Η λογοδοσία, αν ε, δεν υπάρχει και η μάθηση, είναι περιορισμένη λογοδοσία. Δηλαδή μπορείς να πεις τόσοι άνθρωποι καταρδίστηκαν, έλαβαν χώρα τόσες δραστηριότητες σε διάφορα μέρη και δεν μπορείς να πεις τι έχει αλλάξει, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά είναι προβληματικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη συστηματική ανάλυση και κατανόηση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Έχουν απλουστευτεί οι διαδικασίες μεν, όμως το feedback που είχαμε είναι ότι εξακολουθεί να είναι επιθυμητό να υπάρχει μεγαλύτερη απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσο το δυνατόν περισσότερο. Φυσικά μέσα στα όρια των διάφορων κανόνων και κανονισμών. Σίγουρα υπάρχουν ε, πολλές ε, αποδείξεις που μας δείχνουν ότι η Κομισιόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν ξέρουμε πώς τελικά θα εξελιχθεί. Γιατί όπως σας είπα, το IPA2 είναι σε αρχικά στάδια εφαρμογή. και δεν ε, περιμένουμε πολλά αποτελέσματα στο στάδιο αυτό. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το στάδιο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από αυτό που σας είπα. Έτσι λοιπόν τα κύρια συμπεράσματα και πορίσματα μπορεί να αλλάξουν λίγο. Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡ η συντονίστρια κυρία Λύση. Να μας συγχωρείτε, κύριος Λύση. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και κύριοι Ευρωβουλευτές. Κύριε Καλαβέρα, ήθελε να έρθει και ζητεί να την συγχωρέσετε. Αλλά είχε κάποια άλλη υποχρέωση και μου ζήτησε να μιλήσω εγώ στη θέση της για να προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, ήδη οι παρουσιάσεις που έγιναν κάνουν την ζωή μου πιο εύκολη γιατί τα καλύψατε τα περισσότερα. Αλλά για να γυρίσουμε λίγο πίσω, να δούμε τη διαφορά μεταξύ προγραμμάτων αναχώρα και προγραμμάτων που καλύπτουν πολλές χώρες. Δεν είπαμε πολλά για αυτά τα προγράμματα, τα πολλαπλά ούτως υπήν. Είχαμε τις σχετικές ενημερώσεις, αλλά αυτά τα προγράμματα είναι λιγότερο γνωστά, μια που γίνεται διαχείριση από τις Βρυξέλλες. Μιλούμε για το 70% της αρρωγής που παρέχεται. Είναι τα βασικά μέσα για να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες σε τομείς προτεραιότητας. Και ε, υπάρχει διαδρομός διάλογος για ε, τα σχετικά έγγραφα στρατηγικής. Αυτά τα προγράμματα αποτελούν αντικείμενο προετοιμασίας των ίδιων των χωρών. Έτσι συστήνουμε εμείς και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός με τις ανάγκες του κάθε τομέα. Επίσης, θα πρέπει να κρύβονται τα βασικά ζητήματα όπως κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, ε, θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών, ε, μεταρρύθμιση του κράτους, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Αυτά τα προγράμματα πολλαπλής κάλυψης επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως τα IPA και όπως θα θυμάστε στις τελευταίες διαβρύνσεις δεν είχαμε τέτοια και τώρα έχουμε 20-25% κάλυψης της περιφερειακής πολιτικής που αφορά την τωρινή περίοδο διεύρυνσης. Θέλουμε να υπάρξει συμπλήρωση αυτών των προγραμμάτων και οι τομείς παρέμβασης κατονομάζονται εάν υπάρχει ανάγκη για αρρωγή, για κάποια διασυνορικά προγράμματα, για εναρμονισμένες προσεγγίσεις και για διευκόλυνση με εμπειρογνώμονες ή περιφερειακές υποδομές. Πρέπει βέβαια να υπάρχει κάποια συνέπεια μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και αυτών των πολλαπλής κάλυψης προγραμμάτων. Και γι' αυτό γίνονται πολλές συνεδριάσεις και συναντήσεις. Πολλά σημεία επαφή έχουμε και τους ε, συντονιστές των IPA σε κάθε χώρα ε, συναντούμε για αυτά τα πολλαπλής κάλυψης προγράμματα. Και έχουμε τέσσερις άξονες για παρέμβαση σε αυτά τα προγράμματα που καλύπτουν πολλές χώρες για να δούμε εντάχει πρώτα-πρώτα ανατομέα και για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ε, παρέχουμε συμβουλές στις διαφορές χώρες όσον αφορά στην διαμόρφωση των πολιτικών, στις στατιστικές, βελτίωση όσον αφορά τις πολιτικές που χαράσει το κάθε κράτος και έτσι κατελήγουμε σε οικονομίες κλίμακας όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών και έτσι συνεργαζόμαστε με την ε, ε, Παγκοσμία Τράπεζα, το ΔΝΤ, τον νόσα, και χρησιμοποιούμε τα σχετικά ε, χρήματα για οριζόντιες δράσεις όπως το έρασμος ΣΥΝ και πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά την κεντροκατευθυνόμενη λειτουργία της υπόθεσης αυτής. Και βέβαια οι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή βοηθούν στο τι θα γίνει επιτόπου σε κάθε χώρα. Να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει προσοχή ε, στην εκτέλεση των προγραμμάτων και από τα μίντια και από την κοινωνία των πολιτών. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να ισχύει ο κανόνας της, των καλύτερων πρακτικών, υπάρχει περιφερειακή συνεργασία, υπάρχει το σχετικό συμβούλιο που καλύπτεται από το IPA και έτσι προσπαθούμε να βοηθήσουμε την μεταρρύθμιση της λειτουργίας του κράτους, να στηρίξουν το κράτος δικαίου, δίκτυο εισαγγελέων, ε, προσπάθεια καταπολέμησης μέσω αυτού του δικτύου των εισαγγελίων για το, για το οργανωμένο έγκλημα, κατά του δουλεμπορίου, ε, διευκόλυνση του εμπορίου, το ΣΕΦΤΑ, την πλατφόρμα της εκπαίδευσης, και οπότε ε, βοηθούμε σε κάθε επίπεδο. Πολλές χώρες έχουν προβλήματα συνδεσιμότητας, πολύ σημαντικά. Και είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος κατά κεφαλήν ε, για τις επενδύσεις στα Δίκα Βαλκανία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε χρειάζεται συντονισμός. σε σχέση με την περιφερειακή τώρα διάσταση συνεργάζονται με τα IPA και για το περιβάλλον, το κλίμα, την ανταγωνιστικότητα. Το βασικό μέσο ή εργαλείο για τη βοήθεια αφορά το πλαίσιο επενδύσεων. Θα έχετε όλοι ακούσει τον WPIF και αφορά χρήματα από τον κοινωνικό προπολογισμό. αλλά όμως είναι και μια πλατφόρμα για συντονισμό των δωρητών και εδώ συμμετέχει η BRD, IFC και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών. Επίσης, περισσότερα κρατημέλη συμμετέχουν σε αυτήν την πλατφόρμα και έτσι υπάρχει άντληση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παροχή συμβουλών, χρηματοδότηση Επίσης, έχουμε διάφορα ειδικά ταμεία. Ας πούμε για το περιβάλλον, για ανάπτυξη επιχειρήσεων, για διευκόλυνση καινοτομία και βοηθούμε και τις μικροεπιχειρήσεις. Υπάρχει ένα ταμείο για την νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκίνησε για Δυτικά Βαλκάνια και τώρα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή. Να βοηθήσουμε με τα προγράμματα της οργικής συνεργασίας, να υπάρχουν αγαστές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών της περιοχής, αλλά και μεταξύ των τρίτων χωρών της περιοχής. Τι διαπιστώνετε ότι αυτό το πρόγραμμα βοηθά σε συμφιλίωση, σε καλές γειτονικέ σχέσεις. Μα αυτό προσπαθούμε να καταφέρουμε. Με τα προγράμματα που σας ανέφερα. Συνεργασία, εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, συνδεσιμότητα. Μερικά παραδείγματα τώρα. Τα πιο σημαντικά στοιχεία. Δικαιοσύνη, στήριξή της πρωτοβουλίας της κοινωνίας των πολιτών, στήριξη της ποινική δικαιοσύνης, συμφιλίωση, σε επίπεδο στέγασης ε, των εκτοπισμένων. Όσο αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, είναι σημαντικά τα προγράμματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων. γίνεται και η αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων και υπάρχει και ένα θεματολόγιο συνδεσιμότητας. Και εδώ έχουμε στήσει κάποια προγράμματα για δίκτυο μεταφορών, για την ενέργεια και έχουμε και δύο ολάκερες συνθήκες για τη συνεργασία των χωρών της περιοχής. 700 εκατομμύρια ευρώ είναι οι επενδύσεις μας σε ενέργεια και μεταφορές και από χρηματοδότηση IFI έχουμε ε, μαζέψει 2,4 δις. Έχουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα, 83 εκατομμύρια, 69 τις δύο προηγούμενες περιόδους, μικρά προγράμματα. Επίσης έχουμε 9 προγράμματα για τα 9 σύνορα που θέλουμε να καλύψουμε. 1,2 έως 2 εκατομμύρια ετησίως και είναι πολύ δύσκολο να είναι μετρήσιμες οι επιπτώσεις. Αλλά είναι σημαντικό να διαπιστώνετε το ότι στα προγράμματα ΣΥΜΠΙΣΗ υπάρχει ανταπόκριση. Έχουν εμπλακεί και οι τοπικές αρχές. Περισσότερες τοπικές αρχές έχουν κάποιες υπηρεσίες στους Δήμους για την διαχείριση του κοινοτικού χρήματος. Γιατί βέβαια αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προβολή των προσπαθειών τους. Και έχουν εμπλακεί και κάποιοι άλλοι οργανισμοί και οργανώσεις και έτσι εισφέρεται. τη αξία και χωρίς αυτούς το CBC, δηλαδή η διασυνορική συνεργασία, δεν θα γινόταν αυτά τα προγράμματα έχουν ενδυναμωθεί οι δεσμοί όχι μόνο μεταξύ φορέων αλλά και μεταξύ προσώπων στις συνολικές περιοχές. Αλλά έτσι έχουν συσφεχθεί και οι σχέσεις αρχών και κοινωνία των πολιτών σε αυτές τις περιοχές, της διασυνοριακές. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Η την της υπαίθρου, περιβάλλον, πολιτιστικά καλύπτουμε. Έχουμε δίκτυα πολιτιστικά, υπάρχουν πρωτοβουλίες. Είχαμε 37 ε, προγράμματα, έργα 7 εκατομμυρίων για πρωτοβουλίες πολιτιστικές. Πολιτιστικές αξίες, πολιτιστική κληρονομιά. Τον Ιούνιο θα δημοσιεύσουμε ένα δείγμα της σχετικής δουλειάς. Συνεργασία σε επίπεδο τουρισμού. Είναι βασιλική δραστηριότητα αυτή. Σε όλοι έχει ακούσει το Ντινάρικα. Και έτσι προσπαθούμε να έχουμε από Κροατία μέσω Βοσνίας, Μαυροβουνίου ε, ένα μονοπάτι, μια διαδρομή ε, για να αξιοποιηθεί η φυσική ομορφιά της ε, περιοχής. ποιο πρόγραμμα, με ποιο τρόπο θα έχουμε περισσότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που στην αξία. Δεν υπάρχει όμως απάντηση σε αυτό. Αυτά τα πολλαπλά προγράμματα για πολλές χώρες βοηθούν σε εθνικό επίπεδο βοηθούν τις μεταρρυθμίσεις, ε, μάλλον είναι πιο ευέλικτα, πιο γρήγορα αυτά τα προγράμματα, ε, ίσως γιατί έχει αντίστοιχο, έχουν αντίστοιχο ρόλο και οι Βρυξέλλες. Οπότε υπάρχει έτσι ευκολότερη εφαρμογή τους στις ίδιες τις χώρες που καλύπτουν. Πάντως η απάντηση είναι η συμπληρωματικότητα. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να βοηθούν. Και αυτό και εμείς επιδιώκουμε. Να συνεχθούν δηλαδή όλα αυτά με τον πολιτικό διάλογο και σε εθνικό επίπεδο και περιφερειακό. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σήμερα η συνεδρία διεξάγεται γιατί θέλουμε να μάθουμε για ποιο λόγο υπάρχει τόσο περιορισμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν υπάρχει ενίος οικονομικός χώρος, δεν υπάρχουν κοινοί στόχοι, πράγματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για τις χώρες αυτές και που θα προσδώσουν οικονομική ανάπτυξη και ισχύ στις ίδιες αυτές χώρες. Εσεί μου δώσατε μια εξήγηση, τα κονδύλια είναι περιορισμένα. Με αυτήν την διαμεθορική συνεργασία, τι νομίζετε ότι μπορούμε να επιτύχουμε, εκτός από το να γνωριστούν μεταξύ του οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι γνωρίζονται εξάλλου γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια εν μέρη συναποτελούσαν ένα ενίο κράτο. Αλλά γιατί είναι τόσο περιορισμένα τα κονδύλια, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα άλλα ποντάρει σε δημιουργία μεγάλων οικονομικών χώρων και ως ένα βήμα προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να γίνονται δηλαδή συνεργασίες που μετά θα πετύχουν να τι φέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, δόθηκαν λίγα χρήματα στην αρχή για την διασυνορική συνεργασία. Δεν υπήρχε αντίστοιχη δομή στι χώρε. Οπότε ξεκίνησαμε σιγά σιγά, όπως και για τα κράτη-μέλη. Αλλά είπαμε να έχουμε κοινέ ελεκτικές επιτροπές, κοινέ γραμματείες, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε κόσμο, έτσι με το πρώτο είπα. Και είπαμε ότι κάναμε στο ένα, να πάει και στο είπα δύο. Θα σας τα πει και συνάδελφος από το από DG Regio. Οπότε καλύπτουμε και τις χώρες, είπα και τα γειτονικά κράτη. Όσον αφορά τώρα το εμπόριο διασυνοριακά στην περιφέρεια. Αυτό είναι η ψητή προτεραιότητά μας. Έχουμε ένα περιφερειακό κέντρο συνεργασίας για κινητικότητα, διευκόλυνση εμπορίου για την ψηφιοποίηση για τα τελωνιακά θέματα. Αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Και βέβαια ελέγχουμε εάν οι χώρες τηρούν τις υποσχέσεις τους όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν δεσμευτεί να κάνουν. Και μόνο το ότι ξεκίνησε μια τέτοια προσπάθεια αποδεικνύει ότι υπάρχει εμπόριο μεταξύ των χωρών της περιοχής. Και αυξήθηκαν οι εμπορικές ζωές τότε που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Και χτες στο Λονδίνο το είπε ο Πρωθυπουργός της ε, Σερβίας ότι Κίνα, Ρωσία και Τουρκία όλες μαζί έχουν λιγότερες εμπορικές ροές με τη χώρα του, τη Σερβία, από τη Βοσνία. Κύριε Παλαούρα, από την Ελληνική Βουλή. Μικρόφωνο παρακαλούμε, κύριε Παλαούρα. That's right. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων ότι σε σχέση με το κρίσιμο θέμα που συζητάμε σήμερα η θέση μας είναι σταθερή και σαφώς εκπεφρασμένη. Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της έμφασης στη μακροπεριφερειακή συνεργασία σε όλα τα Βαλκάνια με αιχμή τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση διασυνοριακών υποδομών από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα σε αρκετές περιφερειακές συνελεύσεις στις οποίες συμμετέχουμε ως Βουλή, ως Βουλή των Ελλήνων όπως εκείνη της πρωτοβουλίας για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιωνίου αλλά και στην αντίστοιχη που αφορά συνεργασία των χωρών του Ευξήνου Πόντου. Είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης έργων σε περιεθνικό επίπεδο δημιουργεί πράγματι ευνοϊκές συνθήκες περιφερειακής ολοκλήρωσης. Εμπεριέχει όμως και μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις οφειλόμενες και σε ευρύτερα πολιτικά προβλήματα όπως αυτά που ταλαιπωρούν συχνά τα Βαλκάνια. Τα κράτη των Βαλκανίων έχουν ανάγκη από τα μεγάλα διαβαλκανικά έργα και έχουν ευνοηθεί σε κάποιο βαθμό, θα έλεγα αρκετό, αρκετά σημαντικό από όσα έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμή. Παραδείγματο χάρη, ο εξυγχρονισμό του οδικού δικτύου των Δυτικών Βαλκανίων και η ένωσή του με την ελληνική εκνατεία αποτελεί μοκλό σταθερή ανάπτυξη και του ελληνικού τουρισμού. Τα έργα υποδομή σε σχέση με τι διασυνοριακέ εισόδου τη χώρα επίση είναι σημαντικά. Θα πρέπει όμως να δούμε περισσότερα στοιχεία και είναι και πρόταση που θα παρουσιαστεί στις ε, σχέσεις με την ε, Κομισιόν όπως η πύλες εισόδου με την ΦΥΡΟΜ και με την Τουρκία αλλά και η δάτινη ε, συνεργασία με την Ελλάδα και Βουλγαρία γεγονός που πρώτον θα μειώσει τις πλημμύρες και δεύτερον θα δημιουργήσει όρους για την αγροτική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν ανάγκη από κοινέ προσεγγίσεις σε σχέση με τα έργα ανάπτυξη και περιφερειακής συνοχής και αυτό είναι και το κοινό ζητούμενο και σε όλες τις διασκέψεις στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι η μακροϊπεριφερειακή ανάπτυξιακή των Δυτικών Βαλκανίων αποτέλεσε ένα από τα ιδιαίτερα αντικείμενα του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που διοργάνωσε η ελληνική κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη την άνοιξη που μα πέρασε. Ταυτόχρονα και στην τετραμερή διάσεψη Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, στην οποία συμμετείχε πριν από ημέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργό. Μάλιστα εκτές στο Λονδίνο, στη διαδικασία του Βερολίνου, η Ελλάδα κλήθηκε για πρώτη φορά και έγινε τακτικό μέλος σε, ένα, ε, σε μια οργάνωση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για όλα τα Βαλκάνια. Ξαναλέω, η διαδικασία γνωστή ως διαδικασία του Βερολίνου. Θα ήθελα να προχωρήσω και με μία λέξη για την αξία συμπερίληψη στο κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τη συνανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων και της Σερβίας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι κομβικό να ενωθούμε όλοι σε κοινού αναπτυξιακού στόχου, οι οποίοι όχι μόνο θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωή των πολιτών μα, αλλά ταυτόχρονα θα διευρύνουν και τα πεδία κοινωνική σύγκληση που τόσο έχουμε ανάγκη. Μια τέτοια προπτική φαίνεται να ενισχύεται και από την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή μεταξύ Ελλάδας και Φύρων και επίκειται και μια συμφωνία με την Αλβανία που θα βοηθήσει στην οικονομική ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών μεταξύ αυτών των κρατών και της επιχειρηματικότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και ανάπτυξης. Τα Βαλκάνια έχουν μια ιστορία πολύ κακή. Πόλεμοι, ο, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε από τα Βαλκάνια, αντιπαραθέσεις μέχρι πρόσφατα και επομένως πρέπει να δούμε και εθνικισμός φυσικά. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην δει σαν λογιστής τη νέα προσπάθεια ενίσχυσης των Δυτικών Βαλκανίων. Πρέπει να το δούμε μια πολύπλευρη εικόνα. Εικόνα ιστορική, εικόνα που έχει αντιπαραθέσει ακόμα και σήμερα και η οποία όμως βελτιώνεται και πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη βελτίωση. Τα διαθέσιμα εργαλεία αναπτυξιακά ταμεία που ανέφεραν οι συνάδελφοί μου για τις υποδομές, για τα λογίστης, για τις μεταφορές, για την ενέργεια, για την ψηφιακή διακυβέρνηση, πρέπει να, να μπουν και στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα επιμελητήρια, τα εμπορικά επιμελητήρια θα μπουν, θα, μπει, θα ο, ε, η, η ΟΤΑ, δηλαδή η Δήμη και οι περιφέρειες της χώρας, θα μπούμε σε ζητήματα όπως το περιβάλλον. Να σας πω ένα παράδειγμα, το καταλάβετε. Η πρέσπες που έγινε η συνάντηση ε, του Έλληνα Πρωθυπουργού Τσίπρα με τον ομόλογό του της Φίρομ Ζάεφ ήταν στις πρέσπες ένα πανέμορφο μέρος ε, στην περιοχή μας, πανέμορφο μέρος, το οποίο όμως έχει προβλήματα περιβα... περιβαλλοντολογικά. Άρα θα πρέπει να βλέπουμε και τέτοια ζημιά. Και τέλος με το πολιτισμό. Θα βάλουμε τα πανεπιστήμια μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Θα βάλουμε το ενδιαφέρον παιχνίδι, το, το εννοώ σαν στρατηγική. Θα βάλουμε την κοινωνία των πολιτών. Θα δούμε ζητήματα που μας αφορούν όλους και την Ευρώπη την κεντρική αλλά και, τη, και την Ευρώπη προς την πλευρά των Βαλκανίων όπως είναι το προσφυγικό. Είναι καινούρια ζητήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η Βόρεια Ελλάδα, συνάδελφοι, μπορεί να γίνει ατμομηχανή ανάπτυξης και ευρημερίας. Αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καθυστερήσει και να δείξει μεγαλύτερη ζέση. Είπατε κάτι κυρία Πρόεδρε, δεν είναι η προσπάθεια, αν δεν είναι να γνωριστούμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, είναι πολύ καλό πράγμα να γνωριστούμε μεταξύ μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μην καθυστερεί και να δείξει μεγαλύτερη ζέση γιατί τότε το κενό που θα υπάρξει στα Βαλκάνια θα αφαιθεί πλήρως σε άλλα κράτη. Κάτι υπονόησαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Σε άλλες δυνάμεις. Θα τελειώσω με μία φράση που είπε χτες στο Λονδίνο, στη, στην ε, διάσκεψη του Βερολίνου, έτσι λέγεται, η κυρία Μογκερίνη. Η συμφωνία εννοεί Ελλάδας Φύρων είναι έμπνευση για την Ευρώπη. Χρειάζεται όμως διαρκή στήριξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσουμε να ενστερνιστούμε τα θερμά σας λόγια και, τα, και τις προτροπές σας, αλλά δεν είμαστε τίποτα παραπάνω παρά ε, ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Πάντως ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ο κύριος... Όλοι μας να πούμε καλές ε, κουβέντες. Ασφαλώ και θα το κάνουμε. Γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σλοβενικά όμως. Πρόσφατα ήμουν αρκετά αφοσιωμένος στο έργο που γίνεται εντός των χωρών των Νοτικών Βαλκανίων. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συνεδρίαση και που συζητούμε το μέσο προενταξιακής βοήθειας ως το πιο σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής προοπτικής ε, για τις χώρες της περιοχής. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια. Δεν θα πρέπει να μιλάμε εδώ για το κόστος, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε για τις επενδύσεις στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν συζητάμε αυτά τα κονδύλια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιε θα είναι οι στρατηγικές επενδύσεις που θα γίνουν από τα κονδύλια αυτά. Ο προηγούμενο ομιλητή από την Ελλάδα ήδη τόνισε την πτυχή αυτή. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, χρειαζόμαστε καλά αποτελέσματα και διαφάνεια. Και τα δύο είναι ζωτικά για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής προοπτικής ε, στις χώρες της περιοχής. Τώρα, για να μπούμε στις λεπτομέρειες. Θα ήθελα να καλωσορίσω μία από τις παρουσιάσεις που τόνισε ότι οι δικαιτικές διαδικασίες θα πρέπει να πλουστευτούν. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με τη δήλωση αυτή. Αυτό φυσικά ισχύει και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ε, πετύχουμε την απλούστευση των δικαιτικών διαδικασιών, σίγουρα αυτό δεν θα βλάψει στην αύξηση της διαφάνειας. Και τέλος, δεν θέλω εδώ να είμαι ιδιαίτερα διδακτικός. Όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι υποψήφιες χώρες, δεν διαπραγματεύονται μόνο με τις Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει να πείσουν και το κάθε ένα κράτος μέλος ξεχωριστά που μπορεί να έχει διαφοροποιημένες απόψεις για το θέμα. Η δική μου εμπειρία μου λέει ότι όλοι καλωσορίζουν αυτά τα προγράμματα που τονίζουν την επιθυμία για συνεργασία εντός των χωρών, μεταξύ των χωρών, μεταξύ υποψηφίων χωρών και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα τέτοιας συνεργασίας ε, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και τονίζονται γιατί είναι γνωστό ότι υπήρχε πόλωση στην ε, περιοχή στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν η ειλικρινής μου επιθυμία είναι όλοι να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στο να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών αυτών. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Άκερμαν για την λαμπρή παρουσίαση που έκανε και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Πέτερλε για τα ενθαρρυντικά του λόγια για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το σχόλιο μου θα αναφερθεί στην ορατότητα και στα αποτελέσματα και στην έκβαση και θα πω δύο πράγματα. Πρώτο, νομίζω και μιλώ για τη χώρα μου, νομίζω ότι αν μπορέσουμε να αποδώσουμε την συμφωνία που υπέγραψε η Δημοκρατία της Μακεδονίας με τη Βουλγαρία για φιλικές γειτονικές σχέσεις, αν μπορούμε να αποδώσουμε την συμφωνία αυτή στην διαμεθοριακή συνεργασία, νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά ήδη για την ορατότητα της συνεργασίας αυτής. Αν επίσης μπορούμε να αποδώσουμε την ιστορική συμφωνία με την Ελλάδα σε αυτήν την διαμεθοριακή συνεργασία και αυτό θα είναι κάτι το θαυμάσιο που καταφέραμε. Λέχθηκε ότι 83 εκατομμύρια δεν είναι αρκετά. Ασφαλώς δεν είναι αρκετά. Αλλά εάν η CBC, η διαμεθοριακή συνεργασία, μπορεί να αποδώσει έστω και αυτό το 1% στις συμφωνίες που κατάφερε να υπογράψει η χώρα μου με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα θα είναι τεράστια απόδοση. Φανταστείτε τι θα γινόταν εάν τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά αυξηθούν όπως και άλλα κονδύλια για την IPA. Από την άλλη μεριά να πω κάτι άλλο. Κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Για να είναι ορατά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, για να φανούν δηλαδή τα αποτελέσματα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, νομίζω ότι και εσείς και εμείς πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και γρήγορα. Γιατί, διότι άλλες χώρες, είτε μιλούμε τώρα για ανατολικές χώρες ή οποιασδήποτε άλλες από την Μέση Ανατολή, είναι πιο γρήγορες από ότι εσείς και είναι και πιο γρήγορες από ότι εμείς. από την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, θα έλεγα, έχουν καταφέρει αυτές οι χώρες να είναι πιο επιτυχημένες από ότι εμείς με μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστηρίζονται για παραπάνω από 25 χρόνια στη χώρα μου. Και νομίζω ότι αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται κάποιο, κατά κάποιον τρόπο από χώρε τη Μέση Ανατολή ή από χώρε ε, τη Ανατολή, είτε είναι η Ρωσία είτε άλλοι. Μπορώ να σα πω πολύ ειλικρινά ότι οι χώρε αυτέ είναι πλέον πιο επιτυχημένε στα Βαλκάνια από ό,τι οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κονδύλια που διαθέτουν. Είτε λοιπόν μιλούμε για την απλοποίηση, απλούστευση, simplification, είτε για αυτά τα κονδύλια ή για οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, αλλά να δουλέψουμε και με ταχύτητα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτές και να ξεπεράσουμε και αυτή την ας πούμε περιορισμένη ορατότητα των κονδυλίων της Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Ελπίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που προσπαθώ να πω. Αλλά είναι πράγματι σημαντικό. Ο Έλληνας συνάδελφός μου είπε κάτι σημαντικό. Πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα και συμφωνώ απόλυτα και με εσάς ότι ε, έχουμε ανυπομονησία, θέλουμε να μπούμε το δυνατόν ταχύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξάρτητα από το ότι υπάρχουν βεβαίως κάποια κριτήρια που πρέπει να, να ε, πληρωθούν για να μπορέσουμε να, για να μπορέσουμε να ενταχθούμε και εμείς σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Αλλά και εσείς πρέπει να μας πιέσετε για να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Κροατία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί στις 6 έχω μια πολύ σημαντική εκδήλωση αθλητικού χαρακτήρα, όχι πολιτικού χαρακτήρα. Λοιπόν, μιλάμε για τη διασυνορική συνεργασία ως ένα σημαντικό εργαλείο το εργαλείο αυτό χρησιμεύει για την ευαισθητοποίηση των πολιτών προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τα ωφέλη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στη συνεργασία μεταξύ υποψήφιων χωρών και κρατών μελών. Ακόμη και αν τα χρήματα που επενδύονται στη διασυνοριακή συνεργασία αφορούν προγράμματα χαμηλής αξίας, ε, κυρίως ε, ε, υποδομές, αυτά είναι τα πιο ορατά. Αυτά τα project, αυτά τα έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί είναι ορατά σε τοπικό επίπεδο. Η Κροατία είχε πολύ καλή, πολύ καλή εμπειρία ως υποψήφια χώρα στα πλαίσια της συνεργασίας με τη Σλοβενία και την Ουγγαρία. Εγώ προσωπικά συμμετείχα σε προγράμματα CBC με σλοβενικούς δήμους και είχαμε πάρα πολλά διδάγματα, όχι μόνο για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το πώς να είμαστε διαφανείς και το πώς θα καταπολεμούμε τη διαφθορά. Αυτές οι περιβόητες διαδικασίες που δεν αρέσουν συνήθως ε, στους άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι πολύπλοκες, είναι ακριβώς αυτές οι διαδικασίες που κάνουν τους τοπικούς αξιωματούχους ε, να κατανοήσουν ε, πώς λειτουργούν οι δημόσιες συμβάσεις, ε, να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους με σοβαρό τρόπο, τους κάνει να μειώσουν τη διαφθορά σε τοπικό επίπεδο και να αυξηθούν οι επενδύσεις. Όταν μιλάμε για τα προγράμματα σύμπισης στα Δυτικά Βαλκάνια, είναι σημαντικό να πούμε ότι οι καλές ε, σχέσεις γειτονία είναι σημαντικές για να ξεπεραστεί μια δραματική κοινή ιστορία. Και συγκεκριμένα προγράμματα θα καταστήσουν δυνατό να έχουμε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, έτσι ώστε οι πολίτες να δουν ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν πράγματι να βελτιώσουν τη ζωή τους μέσω από συγκεκριμένα προγράμματα στις πόλεις, στα χωριά τους. Θα μπορέσουν έτσι να δουν οι πολίτες ότι είναι καλά τα προγράμματα και με τη σειρά τους οι πολίτες θα κάνουν τις κυβερνήσεις τους να οικοδομήσουν καλύτερες σχέσεις γειτονίας. Και τέλος κάτι που αφορά τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας, τα προγράμματα αδελφοποίησης όπως λέγονται. Ε, Δυτικά Βαλκάνια, η Κροατία έχει τις ικανότητες να ελοπίσει τέτοια προγράμματα. Δεν είναι μόνο ότι μας βοηθά να κατανοήσουμε ε, τους, ε, τους άλλους καλύτερα γιατί έχουμε κοινή γλώσσα. Μπορεί να μάθει κάποιος και κάποια άλλη γλώσσα, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά προερχόμαστε από το ίδιο κράτος, ε, γνωρίζουμε ε, το σύστημα και σημαίνει ότι μπορεί να υποφεληθούμε από τις ίδιες λύσεις. Αλλά καθώς έχουμε μεγάλη πείρα, η Κροατία μπορεί να είναι επικεφαλής του προγράμματος, μπορεί να είναι αρμόδια για το πρόγραμμα, αλλά για να είναι κάποιος αρμόδιος για το πρόγραμμα πρέπει να έχει πολύ πείρα Και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε προγράμματα υψηλής ποιότητας. Και φυσικά αυτά είναι και τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το feedback και για μας. Βεβαίω όλα τα πράγματα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και θα συμφωνήσω σε πολλά πράγματα μαζί σας. Η κυρία Αγγέλοβα από την Βουλγαρία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. This side. It's good now. Αλλάζει μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρώτα πρώτα σας ευχαριστούμε για το ότι διοργανώσατε τη σημερινή συνάντηση. Πρώτα πρώτα να πω ότι βεβαίως πιστεύω ότι η επιτυχής και ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων με τη βοήθεια της Ένωσης ε, είναι κάτι το οποίο θα γίνει εφικτό εάν μπορέσουμε να έχουμε τις κατάλληλες δραστηριότητε και οι επενδύσεις εκεί είναι επενδύσεις προς χάρη της Ευρώπης. Να σε στα βουλγαρικά. Εάν είναι δυνατόν η χώρα, ξέρετε, θέλει διακαώς να συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα διασυνορικής συνεργασίας και έτσι να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε κάποιες εταιρικέ σχέσεις σταθερές, μακρόπνοες με τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στα πλαίσια των προγραμμάτων η χώρα θέλει να καταβάλει προσπάθειες ούτως ώστε να επιληθούν τα κοινά προβλήματα και να βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες να προετοιμαστούν για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για κάθε υποψήφια χώρα. Να εστιαστούμε στην συνδεσιμότητα και την θεία συνδεσιμότητα που είναι πολύ βασική για να πετύχουμε την επιθυμητή ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Να υπάρχει αυτή η περιαφρική συνεργασία, να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων. Επίσης, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Συνεργαζόμαστε μέσω πολλών φορέων και πετυχαίνουμε θετικές συνέργειες. Έχουμε την μακροστρατηγική της Ένωσης για την ε, περιοχή του Δουνάβιος. Στόχος αυτής της μακροστρατηγικής είναι η ολοκλήρωση. Υπάγονται εδώ 14 χώρες. Τρεις από αυτές τις χώρες είναι χώρες Δυτικών Βαλκανίων. τα συμπεράσματα από τη διαδικασία προσχώρηση στην Ένωση κατέδειξαν στο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξει κανείς την ε, περίοδο της μετάβασης από εκεί που είναι υποψήφιο κράτος μέλος να γίνει πλήρες κράτος μέλος. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβλέπονται οι κατάλληλοι πόροι για IPI στο καινούργιο CFP και να υπάρχουν επίσης τα κατάλληλα προγράμματα πλαισίωσης για αμέσως μετά την προσχώρηση. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχή προσχώρηση, όλες, όλα τα προβλήματα, όλες οι προκλήσεις θα πρέπει να έχουν ε, γνωστοποιηθεί στις υποψήφιες χώρες και στα κρατημέλη. Οπότε αυτό είναι καθήκον των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία για τους στρατηγικούς στόχους της προσχώρησης. Επίσης θέλω να σας τονίσω ότι για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εδαφική ολοκλήρωση και καλύτερη ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν διάφορα μέσα και μηχανισμοί θα συνεχίσουν να βοηθούν στην ε, καλή περιφερειακή συνεργασία. Ανάλογα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής που θα γεφυρώσει τις διαφορές. Σας ευχαριστώ πολύ για μια φωνή που ακούστηκε για τις πιο ε, καινούργιες, με τις χώρες που έχουν έρθει πιο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε. Ευχαριστώ. Προέρχομαι από τη Σερβία και λέγομαι Κόμιτς. Όσο σύντομο μπορεί να προσπαθήσει να είναι οποιοδήποτε βουλευτής, θα προσπαθήσω να μοιραστώ μαζί σας το πώς από κοινού μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε την ε, καλύτερη απάντηση στην προφανή ερώτηση εδώ. Δηλαδή, η αξία των χρημάτων που δίνεται από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους στην περιοχή μας. Αξίζει τον κόπο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όταν ε, βλέπω τους δημοσιονομικούς ελέγχους ε, στη Σερβία, και πολλά έχουν γίνει, κατόπιν ε, μπορώ να πω ότι υπάρχουν φορείς για την καταπολέμηση της ε, ευεξαίρεσης ε, και κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ε, υπάρχει γενικά βελτίωση στην προσέγγιση της πολιτικής της που επικεντρώνεται σε περιφερειακή συνεργασία για την επίλυση πολύ δύσκολων ιστορικών ζητημάτων στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά όμως, το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει τόσο λίγη συνεργασία. Όταν δίνονται χρήματα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, γιατί αυτά τα κονδύλια δεν παράγουν περισσότερη συνεργασία και ζω στην περιοχή και μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, πέρα από τον να αυτό το απλό. Θα σας πω και κάτι ειλικρινές, γιατί διστάζουμε να αναλάβουμε το μέλλον μας. Διστάζουμε να γίνουμε οι κύριοι της περιοχής. Προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας, λαμβάνοντα υπόψη ο ένας τον άλλο και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εκεί για να επιβάλλει λύσεις για μας. Γιατί τίνουμε να σας λέμε ψέματα, πιστεύουμε ότι είστε πιο έξυπνοι και πιο όμορφοι από εμά. Και γιατί δεν πραγματικά αναλαμβάνουμε την κυριότητα της περιοχής. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων κοινών εντός της περιφέρειας που αντικατορίζονται στην ευφύ σε ερώτηση γιατί τόσο λίγη συνεργασία ενώ υπάρχουν τόσο πολλά χρήματα που οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι είναι έτοιμοι να μοιραστούν μαζί μα για τη βελτίωση τη συνορική συνεργασία, για τεχνική βοήθεια, για να βοηθήσουν του ανθρώπου προσωπικά να επενδύσουν σε σχολεία, στην εκπαίδευση, στην υγεία. Όμως, το δεύτερο μέρος της απάντησης αυτής είναι ότι και εμείς ίδιοι δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση. Αν γίνει κάτι τέτοιο, αν υπάρχει βελτίωση και βούληση για συνεργασία και αν υπάρχουν ε, οι καταληφορείς ε, εποπτείας, γιατί αυτό δεν είναι δημοφιλές και δεν είναι ορατό. Γιατί δεν ε, λαμβάνεις μια απάντηση στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να χάρη στη Σερβία και λένε ότι η Ρωσία επενδύει η Ρωσία δεν επενδύει ένα ευρώ. Όμως η αντίληψη των ανθρώπων δεν συνάδει με τα κονδύλια που λαμβάνουμε από εδώ, που πραγματικά τα δαπανούμε σωστά και τα διαχειριζόμαστε σωστά. Δεν μιλάω εδώ τώρα για την ε, κατάχρηση κάποιων κονδύλιων εδώ και εκεί. Συμβαίνει αυτό, το γνωρίζουμε. Τελικά η δική μου ανησυχία είναι γιατί δεν είμαστε αρκετά γενναίοι για να αναλάβουμε την κυριότητα του τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Γιατί χρειαζόμαστε διαμεσολαβητές στις συνεδριάσεις μας, είτε πρόκειται για την υπηρεσία εξωτερική δράσης, είτε τα έρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί μας, που θέλουν πράγματι να μας βοηθήσουν να ξοδέψουν χρόνο και να αναπτυχθούμε νωρίτερα σε σχέση με το τι θα κάναμε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ποτέ δεν θα σταματήσω να πιστεύω στις ε, αξίες και στην ομορφιά των ευρωπαϊκών ιδεών. Και θα θέλαμε να δούμε περισσότερους ε, Ευρωπαίους να το θυμούνται αυτό και να εναγκαλίσουν την ε, καρδιά της ευρωπαϊκής ιδέας. Αυτό είναι ένα σχέδιο ειρηνευτικό. Στην περιοχή έχουμε μια επιτυχία. Δεν θα συνέβαινε χωρίς τις ευρωπαϊκές ιδέες. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ζωντανό στην περιοχή. Και δεν το βλέπω τόσο έντονα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί βλέπω ότι αυτό συνδέεται με το πώς ε, η χρηματοδότηση που μπαίνει στην περιοχή μπορεί να δαπανηθεί με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Και πώς εσείς, ε, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς που εργαζόμαστε από μόνοι μα. όταν θα γίνουμε μέλος μπορούμε να πούμε αυτό οφείλεται στο ότι εσείς δώσατε τα χρήματα των φορολογουμένων και ήταν πολύ καλό που δόθηκαν στην περιοχή μας αλλά δεν πρόκειται περί χρημάτων. Αυτή είναι μια ιδέα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας με την ελπίδα ότι θα έρθει και η στιγμή αποπληρωμής από την περιοχή και τώρα εμείς πρέπει να αποδείξουμε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποδείξουμε ότι άξιζε να πιστεύετε σε εμά, να επενδύετε στους ανθρώπους και ότι είναι καλό να επενδύουμε μαζί στο κοινό μας μέλλον. Όποτε έλθει αυτό το μέλλον, θα έλθει. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Μένει ακόμα μία, ε, μία συνάδελφος που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Οι διερμηνείς μας ε, καταθέτουν τα όπλα ακριβώς στις 18 και 30, θέλω να πω δηλαδή, πάβουν την εργασία τους. Εξημών ποιος καταλαβαίνει αγγλικά. Ποιο μάλλον δεν καταλαβαίνει αγγλικά, ποιο δεν καταλαβαίνει αγγλικά από του προσκεκλημένου μα από τι χώρε ε, των Βαλκανίων. Ποιο δεν καταλαβαίνει αγγλικά. Όλοι καταλαβαίνετε αγγλικά. Διότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά από την αποχώρηση των διερμηνών στι 18 και 30 στην αγγλική γλώσσα. Ο κύριο Βούκιτ ακολουθεί από το Μαυροβούνιο. You can still speak in your language. Μπορείτε, μπορείτε ακόμη να μιλήσετε στην γλώσσα σας μέχρι τις 6.30 όμως. Σα Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ο κ. Φούτσης. Δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω τη γλώσσα από την οποία προέρχομαι, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου. Και οι φίλοι των γειτονικών χωρών της περιοχής μας θα συμφωνούν ότι το Μαυροβούνιο είναι χώρα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από πολλές απόψεις. Και επί Ιουγκοσλαβίας είχαμε τις ίδιες ιδιοτυπίες. Η πιο μικρή χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Πρώτα-πρώτα λέει ο κύριος Βούκοβιτς. Και έχουμε 600.000 κατοίκους, σήμερα με την τελευταία απογραφή, πάντως έχουμε και μετανάστες. Ε, οπότε πάμε στις 600.000 ε, και λίγο πιο κάτω. Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μειονέκτημα όσον αφορά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρσι ε, γίναμε μέλος του ΝΑΤΟ. Είχαμε τα πιο πολλά κεφάλαια από οποιαδήποτε άλλη υποψήφια χώρα. Τώρα είμαστε στην φάση ολοκλήρωση του κλεισίματος των κεφαλαίων 23 και 24 κάνουμε μεγάλη πρόοδο σε αυτό το μέτωπο και επίση ε, προσπαθούμε και στον τομέα της διασυνορικής εργασίας. Οι γείτονε μας εκτός από την Κροατία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίση την Αδριατική που μας ε, χωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία που είναι απέναντι την άλλη μεριά. Οπότε, για να μπορέσουμε να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περάσουμε, να παρακάμψουμε τους γειτονές μας. Τι να κάνουμε επομένως εμείς οι Μαυροδονοί. Πρώτα-πρώτα διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια επιβράδυνση του ρυθμού προσέγγισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για τα κονδύλια, για τους πόρους. Έχουμε απορροφήσει χρηματοδότηση και θα δούμε κατά πόσο πιάσαν τόπο αυτά τα χρήματα. Και η ώρα της αλήθειας είναι όταν γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντως όπως και να έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλιώς είναι άδικο. Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε Σερβία με Μαυροβούνιο. Η Σερβία είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Με την Βοσνία που είναι τρεις φορές πιο μεγάλη, ούτε με τη Βοσνία μπορούμε να συγκριθούμε για τα κριτήρια. Κάποια θεσμικά όργανα της Ένωσης λένε ότι πληρούμε όλα τα δυναμικά κριτήρια όσον αφορά την ένταξή μας στην Ενεργειακή Ένωση για φυσικό αέριο, για ενέργεια κλπ. Οπότε συνεχίζουμε την προσπάθεια να κλείσουμε τα κεφάλαια 23 και 24. Είναι προκειμένου θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα. Βέβαια κατά συνεχεία αλλάζει, ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κλείσαμε, τελειώσαμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε το έργο μας. Υπάρχει και το θέμα της διαφθοράς, υπάρχει το θέμα ε, του οργανωμένου εγκλήματος και αν προσπαθήσουμε να, αποτιμήσουμε ποσοτικά αυτά τα κεφάλαια, ε, θα δούμε πόσο δύσκολα είναι αυτά τα κεφάλαια για μας, για να τα κλείσουμε. Οπότε, φυσικά και είναι πρωταρχική σημασία οι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε χωρίς την ε, χρηματοδότηση αυτή. Και για το εξωτερικό εμπόριο, ε, όλες οι χώρες Βαλκάνια είναι ελληματικές όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο. Επίσης έχουμε χρέος το οποίο είναι πάνω από τα κριτήρια του Μάστιχ, το 60%. Είναι και το θέμα τώρα της ε, Ευρωζώνης, των χωρών που έχουν το ευρώ. Εμείς δεν έχουμε, επομένω δεν έχουμε νομισματική πολιτική. Ούτε πολιτική άμυνας. τα λάθη είναι δική μας ε, ευθύνη όπως επίσης και το ότι εξαρτώμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση την πιο μεγάλη δύναμη στρατιωτική και οικονομική. Οπότε το δικό μας μήνυμα ποιο είναι. Θα πρέπει με αφορμή αυτήν τη συνάντηση να προβληματιστούμε να κάνουμε την διαφορά. Είναι μέσω των όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ξαναλέω ότι θα είναι χρήσιμο να συνεργαστείτε όλοι μεταξύ σας πολύ στενότερα και να δείξετε μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας. Θα δώσει και σε εμάς την αίσθηση ότι και η ένταξη θα είναι επιτυχημένη. Η Ένωση πρέπει να είναι ένα πρότυπο επιτυχίας και για σας πρότυπο επιτυχίας και είναι βασισμένη στη συνεργασία. Δεν μπορεί το, το πρότυπό σα να είναι ότι η Ευρώπη θα έρθει και θα σα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι αδυνατόν. Κύριε Πόλοβα, να σας δώσω το λόγο για το θέμα των έργων, της ορατότητα και τη συνεργασία. Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε. Okay, good afternoon, uh, Mrs. Καλό σας απόγευμα, κυρία Γκρέσλε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αξιότιμα μέλη των ε, κρατών μελών και των δικαιούχων του Μέσου Πρωτοεξιακής Βοήθειας. Ε, μου ζητήθηκε σήμερα να μιλήσω για την προβολή και την αποτελεσματικότητα του Μέσου Πρωτοεξιακής Βοήθειας και τη διασυνοριακή συνεργασία με τα κράτη-μέλη εδώ μέχρι τώρα. Ακούσαμε να γίνεται μεγάλη συζήτηση για το θέμα της συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια μεταξύ των ίδιων των χωρών. Επομένως, θέλω να αποσαφηνίσω ότι έχουμε δύο είδη προγραμμάτων. Το ένα είναι, είπα, είπα μεταξύ δηλαδή των χωρών, αυτών καθ' αυτών, και το άλλο είναι μεταξύ των δικαιούχων, είπα, και των κρατών μελών. τα προγράμματα αυτά, για τα προγράμματα αυτά είναι αρμόδια η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρίτζιο. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για την αποτελεσματικότητα, την ορατότητα, την προβολή και υπήρχε και μια ερώτηση για τη συνεργασία με την Τουρκία. Να ξεκινήσω με το πλαίσιο αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, να υπενθυμίσω τους γενικούς στόχους των προγραμμάτων πράγματι καλύπτουν τα προγράμματα αυτά ή συνεισφέρουν και στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές πολιτικές δηλαδή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή ε, εδαφική συνεργασία που είναι μέρος της πολιτικής συνοχής. Αποτελεί λοιπόν συνδυασμό της εσωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής διεύρυνσης. Εδώ στη διαφάνεια βλέπετε τις επικράτειες που καλύπτονται από τα 10 προγράμματα διασυνορικής συνεργασίας στην περιοχή. Βλέπετε ότι οι επικράτειες που καλύπτονται είναι πράγματι τα Nats 3, δηλαδή οι μικρότερες περιοχές πάνω στα ίδια τα σύνορα. Αυτό επιτρέπει για συγκέντρωση και εστίαση στις ανάγκες στα σύνορα και στη δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τον κατάλογο των προγραμμάτων με τα κονδύλια. Τα κονδύλια προέρχονται και από την χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής και από τη χρηματοδότηση του μέσου πρωταξικής βοήθειας και έχουμε ίσο μερίδιο για κάθε ένα από τα προγράμματα. Βλέπετε ότι το, σε σχέση με το, σε χώρες, είπα, είπα, εδώ έχουμε διαφορετικούς ε, προϋπολογισμούς σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στα ίδια τα προγράμματα, κάτι που θα πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που είναι πολύ σημαντικό είναι η διακυβέρνηση και τα κριτήρια να υλοποιηθεί η συνεργασία συγκεκριμένα προκειμένου ένα διασυνοριακό πρόγραμμα να υλοποιηθεί θα πρέπει πάντοτε να έχουμε εταίρους τουλάχιστον από δύο χώρες και από τις δύο πλευρές των συνόρων μια από συμμετοχή δηλαδή ενός κράτους μέλους και μια συμμετοχή μη κράτους μέλους προκειμένου να ελοπιθεί ένα πρόγραμμα από κοινού. Και μεταξύ αυτής της σύμπραξης θα πρέπει να υπάρχει και ένας εταίρος που θα θεωρείται ε, επικεφαλής εταίρος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα στο σύνολό του και μπορεί να προέρχεται είτε από τα κρατημήλη είτε από μία μη ε, χώρα, μια χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν η κοινωνία των πολιτών, η τοπική αυτοδίκηση, οι τοπικοί φορείς μπορούν να συνεργαστούν με τα κράτη-μέλη είτε με άλλους τοπικούς φορείς είτε με την τοπική αυτοδίκηση εντός των κρατών μελών, σε ισότιμες συνθήκες και μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένα project. Ένα άλλο στοιχείο της αποτελεσματικότητας που αποκαλούμε πλαίσιο επιδόσεων επίσης είναι ενσωματωμένο στον κανονισμό της πολιτικής συνοχής, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων που ισχύει ως αναφορά σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό το χαρακτηριστικό διασφαλίζει ότι στην έναρξη των προγραμμάτων υπάρχουν δείκτες ε, που τίθενται για τις αποδόσεις και για τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρο το τι πρέπει να πετύχουν ε, αυτά τα προγράμματα στο τέλος της εφαρμογής ε, και οικονομική στόχη και ρεαλιστική στόχοι και ελέγχεται η επίδεση των προγραμματών αυτών δύο φορές. Στο μέσο της προγραμματικής περίοδου, το 2019, Έχουμε δηλαδή αυτό το εγχείρημα του χρόνου, όπου θα εξετάσουμε πού βρίσκονται τα προγράμματα σε σχέση με αυτά τα ορόσημα και στο τέλος του προγράμματος, των προγραμμάτων που θα είναι το 2023, πάλι θα εξετάσουμε πώς προχώρησαν τα προγράμματα και αν πέτυχαν τους στόχους που είχαν θέσει υπάρχουν για κάποιες πιθανές κυρώσεις ε, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Φυσικά κανένας ε, δεν ε, θέλει να χάσουν τη χρηματοδότηση τα προγράμματα. Δηλαδή ο κανόνας ε, της ε, των κονδυλίων είναι, αλλά μπορεί να υπάρξουν τέτοιες κυρώσεις, μπορεί να υπάρξουν κάποιοι κανόνες διόρθωσης. Θα ήθελα να κάνω και μία παρέθεση από την ενδιάμεση εξυλλόγηση του ΙΠΑ 2. Έχει γίνει μια αναφορά στην προσθεμένη αξία των προγραμμάτων. Εδώ επαναλαμβάνεται αυτό και δεν νομίζω ότι κανένα στην αίθουσα μπορεί να αμφισβητήσει ότι η διασυνοριακή συνεργασία έχει μοναδική προσθεμένη αξία γιατί κάνει άλλος δεν χρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα και αυτά τα έργα. Τώρα, να στραφώ στα θέματα που αφορούν την προβολή, την ορατότητα. Τα προγράμματα αυτά είναι υπό κοινή διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν υποχρεώσεις και για τους κράτη-μέλη, τις διαχειριστικές αρχές, τα ίδια τα προγράμματα και την Κομισιόν. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουν ε, οι αρχές, ε, αυτό είναι ενσωματωμένο στον κανονισμό, θα πρέπει να υπάρχουν ε, στρατηγικές επικοινωνίας και σχέδια επικοινωνίας για όλα τα προγράμματα, θα πρέπει να συστήσουν ένα μοναδικό, μια μοναδική ιστοσελίδα ή μια πύλη στο, στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός από τα προγράμματα. Νομίζω ότι είναι μια θέα της Ελλάδας από την ε, Φύρο. Και εδώ έχουμε την ιστοσελίδα που μπορείτε να βρείτε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Ένα άλλο παράδειγμα ενός μιας εκδήλωσης προβολής είναι αυτό που λέμε η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Αυτό αναπτύχθηκε από ένα πρόγραμμα που βοηθά τη λειτουργία όλων αυτών των προγραμμάτων, πρόγραμμα Interact, στις 21 Σεπτεμβρίου σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στις χώρες της διεύρυνσης υπάρχουν ε, εκδηλώσεις ε, και τα προγράμματα παρουσιάζουν τι έχουν πετύχει, οργανώνονται εκδηλώσεις από τα προγράμματα, προκειμένου οι πολίτες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνειδητοποιήσουν τι επιτυγχάνεται. Και θα ήθελα να σας καλέσω να παραβρεθείτε σε αυτές τις εκδηλώσεις γιατί πράγματι πάντοτε είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Και ίσως ε, αν έχουμε χρόνο μπορούμε να δούμε και το βίντεο για την Ευρωπαϊκή μέρα συνεργασίας και έχει χρησιμοποιηθεί από τα περισσότερα προγράμματα. Τώρα, από την πλευρά της Κομισιόν θα σας πω τι κάνουμε εμείς ε, για να προωθήσουμε την προβολή των προγραμμάτων αυτών. Μπορεί να ακούσατε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πόλεων ε, και Περιοχών. Είναι το μεγαλύτερη εκδήλωση πολιτικής παγκοσμίω. Ε, συνήθως έχουμε 6.000 συμμετέχοντες, πάνω από 100 εκδηλώσεις, workshops, σεμινάρια και ε, κάθε χρόνο έχουμε ένα σεμινάριο για τα προγράμματα της διασυνοριακής συνεργασίας ε, του Μέσου Προταξικής Βοήθειας ε, και μπορεί να ξέρετε ότι έχουμε δημοσιεύσει τις προτάσεις για τη νέα πολιτική συνοχής όπου έχουμε το νέο κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία όπου θα περιλαμβάνεται και η συνεργασία για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα της απλούστευσης που έχει αναφερθεί εδώ. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, όχι μόνο για την προβολή, αλλά και για τις επιδόσεις, είναι το η πύλη της ανοιχτής ημέρα. Ε, λοιπόν, λυπάμαστε που θα, την ερμηνεία θα πρέπει να σταματήσει εδώ την προγραμματισμένη ώρα λήξης της συνεδρίασης. Per program, what kind of, uh, how is the program uh, progressing? You can see the, the what is planned in terms of, uh, of the uh, investment. You can see what is the progress in the spending as well. If you click on, on any of these